Euh, Καλημέρα σας. Να αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας ε, της Επιτροπής Ανάπτυξης με τις ψηφοφορίες. Θα ήθελα να σας ζητήσω να ε, βγάλετε τις κάρτες ψηφοφορίες σας, ψηφοφορίες σας για να βεβαιωθούμε ότι δουλεύουν ε, οι μηχανές. Άρχιτι ψηφοφορία. Α, εγώ δεν ψήφισα, λέει η πρόεδρος. Πέρα τη ψηφοφορία. Πολύ ωραία, δουλεύει το μηχάνημα. Περνάμε λοιπόν στην ε, ψηφοφορία. Για το έρασμος για όλους, τροπολογία 25, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ, 34 συγγνώμη, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ κατά απόχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται.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 αποχές εγκρίνεται. Όχι, απορρίπτεται, λέει η Πρόεδρος. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικώς. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 32. Κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο της γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Le Πέρας. Εγκρίνεται ομοφόνος. Alors, félicitations, euh, à notre... Συγχαρητήρια στον εισηγητή για την πάρα πολύ καλή έκθεσή του. Περνάμε τώρα στην έκθεση Νέβα. Δεν υπάρχουν τροπολογίες, οπότε θέτω σε ψηφοφορία τη γνωμοδότηση ως έχει. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικός. Πέρας. Εγκρίνεται ομοφόνος. Περνάμε τώρα στην έκθεση του κυρίου Σφένσον για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 3, καταπίπτει. Α. Τροπολογία 3, την ψηφίζουμε τελικά, υπέρ, κατά, αποχές,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 απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική υπαριθμών 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήταν όμως κατά τμήματα ψηφοφορία, οπότε το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 23. Υπέρ, κατά, αποχές, καλύτερα να Ψηφίσουμε ηλεκτρονικός Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 20, 24. Απορρίπτεται λοιπόν. Τέλο πάντων, ισοπαλίας είναι ένας ψήφος, μία ψήφος κατά, 24 λοιπόν υπέρ, κατά, απόχέ. ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Εσείς ψηφίζετε υπέρ ή κατά που δεν έχετε την κάρτα σας. Απορρίπτεται τότε. Τροπολογία 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο της γνωμοδότησης, όπως τροποποιήθηκε, ηλεκτρονικός, άρχεται η ψηφοφορία. Le Πέρας. Εγκρίνεται. Ομοφόνος. Συγχαρητήρια κυρία Βένσον. Ψηφίζουμε τώρα την έκθεση του κυρίου Νόισερ ε, για την εργασία της ε, κοινοβουλευτικής συνέλευσης ΑΚΙ Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροπολογία 1, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3, υπέρ. Κατά,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 αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 4, υπέρ, συγγνώμη, συγγνώμη. Εγώ διαφωνώ με αυτή την προφορική τροπολογία και ο λόγο ε, αυτό έχει εξηγηθεί ε, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρωπαϊκή Ένωση ε,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 κατά αποχές εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε τώρα το σύνολο. Άρχεται η ψηφοφορία. Euh, Μας λείπει μία ψήφος. Πέρας. Εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε τώρα. Τη δική μου έκθεση. Για την επισητιστική βοήθεια. Τροπολογία 1. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τρία υπέρ ε, κατά τμήματα ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος στις 7 άρχεται η ψηφοφορία Le Πέρασε. Εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία για την παράγραφο 2 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικώς την προφορική τροπολογία για την παράγραφο 2 του ΕΛΚ άρχεται η ψηφοφορία Λοιπόν, Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. 18. Συγγνώμη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19. Κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Α, θέλετε να επαληθεύσουμε 23. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τροπολογία 23. Πέρας. Απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 26, τμηματική πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την, την ε, γνώμη όπως έχει τροποποιηθεί. Αρχίζει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ομοφόνος. Merci. Euh, Ψηφίζουμε τώρα. Την έκθεση Μέισνερ για την αλληλευτική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γρυλανδίας και Δανίας. Καμία τροπολογία. Ψηφίζουμε λοιπόν την γνωμοδότηση ηλεκτρονικά παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Le vote est clos. Adopté. Εγκρίνεται με τρεις αποχές. Et voilà. Nous avons terminé Τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες και σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε μισή ώρα στη διάθεσή μας γιατί έληξαν οι ψηφοφορίες νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Οι εμπειρογνώμονες είναι παρόντες. Προχωρήσαμε τάχιστα με την ψηφοφορία μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, τόσο γρήγορα κάναμε τις ψηφοφορίες, κερδίσαμε χρόνο. Αλλά δεν έχουν έρθει οι πυρογνωμονές μας για την ακρόαση, δυστυχώς, οπότε πρέπει να διακόψω για 15 λεπτά. Στις 10 παρατέταρτο θα ξαναρχίσουμε.

η δική μου Thank

δεν

Υπότιτλοι AUTHORWAVE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

Euh, Να ξαναρχίσουμε τις εργασίες μας. Περνάμε στην ακρόαση για την ε, εξασφάλιση των γεών ε, στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες. Η Κατρίν Γκρέζ είναι υπεύθυνη για την οργάνωση του, της ε, ακρόασης για την ε, πειρατεία. Ε, σήμερα αρχίζουμε λοιπόν μια νέα ακρόαση που αφορά την συσσόρευση των γεών ε, στις χώρες τις αναπτυσσόμενες. Θα ε, θέλουμε λοιπόν εμείς να υπάρχει μια εξασφάλιση της έγκαιση ιδιοκτησίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα ήθελα να ε, σας ε, παρουσιάσω την κυρία Στρίφλερ που είναι συνδιοργανώτρια, ο κύριος Κοζούσνικ και ο κύριος Μίτσελ. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συναδέλφους για τη δουλειά τους και τη συνεργασία τους κατά την οργάνωση της ε, ακρόασης. Θα είναι ε, συντονιστές της συζήτησης κατά τη διάρκεια της ακρόασης. Θα περάσουμε στην εξέταση διαφόρων ε, τρόπων ιδιοκτησίας γης στις αναπτυσσόμενες χώρες και μετά θα γίνει μια συζήτηση για το ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην γεωργία. Ε, προκειμένου να επιβιώσει ο ντόπιο πληθυσμό. Θα ε, ολοκληρώσουμε με ανταλλαγή απόψεων για την, ε, με την Επιτροπή και του εμπειρογνώμονε για το πώ μπορούμε τα δικαιώματα τη εγγύου ιδιοκτησία να τα εξασφαλίσουμε και να δούμε τι μέσα υπάρχουν στη διάθεση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορούμε να συνεχίζουμε την προσπάθειά μα αυτή. Η καταπολέμηση τη ισόρρευση των γεών και η εξασφάλιση τη εγγύου ιδιοκτησία είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, και είναι πάρα πολύ σημαντική λόγω της δημογραφικής ανάπτυξης, ε, της αστικοποίησης, ε, μαζικό φαινόμενο στις αναπτυσσόμενες χώρες και στην κούρσα για τις καλλιεργήσιμες γεές μεταξύ των κυβερνήσεων και των πολιτών. Ε, θέλουμε να προστατεύσουμε περισσότερο τους πληθυσμούς αυτούς και ε, εκτιμάται ότι 200 εκατομμύρια εκτάρια γεών ε, υπέστησαν διεθνείς επενδύσεις μεγάλης κλίμακας. Μιλάμε για 200 εκατομμύρια εκτάρια σε 10 χρόνια πάρα πολλοί γεωργοί, κυρίως ε, μικροί γεωργοί μικρών εκμεταλλεύσεων, έχουν χάσει τη γη τους και την ε, ε, επισητιστική τους ασφάλεια, απειλούνται. Τα, τα δύο τρίτα των γέων αυτών ε, αγροκαύσιμα σκοπό έχουν να παράγουν με αποτέλεσμα μεγάλη επισητιστική απειλή. Ε, υπάρχει έκθεση της Oxfam ε, από την 4η Οκτωβρίου ε, που δείχνει ότι η συνολική έκτωση, συνολικη εδώ και 10 χρόνια επενδύσεων καλλιεργήσιμων γεών θα έδινε τη δυνατότητα ένα δισεκατομμύριο άτομα να, να τραφούν που σημαίνει τον αριθμό των ατόμων που πλήττονται από πείνα. Στην Καμπότζη οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις εκτιμούν ε, ότι το 53 έως 62% των ε, αρρώσιμων γεών ε, έχουν χαθεί λόγω ιδιωτικών συμφερόντων. 2003, 20 χρόνια πολέμου, 30% των γεών ήταν τμήμα συναλλαγών εγγύου ιδιοκτησίας μόνο σε 5 χρόνια, εντός 5 ετών. Η συσσόρευση των γεών ε, ενισχύθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε οι συναλλαγές εγγύου διοκτησίας τριπλασιάστηκαν ε, κατά την επισητιστική κρίση του 2008 και 2009. Αυτό με οδηγεί στο να επανεπισημάνω την αναγκαιότητα ε, ε, διευθέτησης ε, των οικονομικών. Ξέρετε όμως ότι αυτό είναι μια τεράστια αποτυχία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλύτερη νομοθεσία λοιπόν για την έγκυο ιδιοκτησία θα ήταν εποφελής για την αποθάρρυνση της διαφθοράς στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω έγκρισης κανόνων υποχρεωτικών για διαδικασίες διαφανής. Δεν λέω ότι πρέπει να εξαγάγουμε το δικό μας μοντέλο σε αλλά το να μεταφέρουμε την τεχνογνωσία μας είναι καλή πρακτική ε, μέσω της αναπτυξιακής συνεργασίας. Η επεξεργασία των πολιτικών ε, της Ένωσης επηρεάζει το θέμα ε, της εγγύου ιδιοκτησίας σε διεθνές επίπεδο. και η, τράπεζα, η Παγκόσμια Τράπεζα έχει ε, μεγάλο ρόλο. Η Oxfam λέει ότι από το 2008 20.000 καταγγελίες υπάρχουν ε, ε, σε διεθνές επίπεδο που λένε ότι τα η Παγκόσμια Τράπεζα συμμετέχει σε σχέδια τα οποία πλήττουν την έγκυο διοκτησία των αναπτυσσομένων χωρών. Πρέπει να στείλουμε λοιπόν ένα ηχηρό μήνυμα για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Ε, ελπίζω ότι η ακρόαση αυτή θα μας δώσει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε καλύτερα τις συνέπειες που οι, διάφορες, ε, οι διάφοροι τρόποι ε, εγγύου ιδιοκτησίας μπορεί να έχει για τη μείωση της φτώχειας και την, ανάπτυξη, την περαιτέρω ανάπτυξη των αναπτυσσομένων χωρών. Ελπίζουμε επίσης να φανεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πρέπει να γίνει μια αναδιάρθρωση μέσω διαφανούς νομοθεσίας που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα των τόπιων πληθυσμών ε, και να συνεισφέρουμε με αυτόν τον τρόπο στην ε, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών αυτών, όπως επίσης και στην επιστημιστική τους ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εποφελούμαστε από ένα πάνελ εμπειρογνωμόνων ε, σημαντικών προσωπικότητων. Να τους καλωσορίσω λοιπόν και θα σας τους παρουσιάσει, θα τους παρουσιάσουν οι συνάδελφοί μας, οι διοργανωτές της ε, ακρόασης. Πρώτα θα μιλήσει η κυρία Στρίφλερ που είναι η συντονίστρια της συζήτησης για το πρώτο τμήμα της ακρόασης αυτής. Σας καλημερίζω όλους. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι μαζί σας σήμερα για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Το θέμα της εγγύου ιδιοκτησίας είναι πολύ σημαντικό μας ενδιαφέρει η πρόσβαση στη γη και η φυσική πόρη. Πρόκειται για ένα σημαντικό διακύβευμα οικονομικό και πολιτικό, διότι ορίζει τα δικαιώματα επί της γης και τον τρόπο κατανομής γεών. Την πολιτική εγκύου ιδιοκτησίας, που φυσικά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Μας ενδιαφέρει η έκθεση Τάις Μπέρμαν, για το μέσο συνεργασίας και ανάπτυξης 14-20 και πολλά έχουν εγκριθεί μέσα στα πλαίσια της αναπτυξιακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει ασφάλεια γεών ανά τον κόσμο μέσα στα πλαίσια σειράξεων και κλειδονισμών οι δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις επενδύουν κατά ένα δις εκτάρια στην Αφρική, Ασία και Λατινική Αμερική για να παράγουν τρόφιμα και βιοκαύσιμα. Αυτό που έχει λοιπόν σημασία είναι να γίνουν επενδύσεις για να υπάρχει καλύτερη αγροτική και διατροφική ασφάλεια χωρίς να πλήττουμε τους αυτόχθονες και τις αυτόχθονες κοινότητες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι χώρες του Νότου θα πρέπει να προβούν στη σύσταση μιας πολιτικής υπέρ των γεών, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική, κοινωνική και θεσμική κατάσταση που αφορά την κάθε χώρα χωριστά. Στόχος είναι να διασφαλίσουμε τη χρήση των γεών με βάση κάθε είδους νομιμότητα, να προωθήσουμε τις οικονομικές πολιτικές οι οποίες να είναι δίκαιες. Πρόκειται για κάτι το πολύ δύσκολο. Μπορούμε να βασιστούμε στο δίκαιο το οποίο μπορεί να είναι και θυμικό δίκαιο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει νομική αναγνώριση, αλλού όμως όχι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι υπάρχει και συλλογική ιδιοκτησία σε ορισμένα σημεία της γης. Θα πρέπει λοιπόν να ορίσουμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των γεών. Ο κύριος Αμπτουλάγε Χαρίσου είναι πρόεδρος ομάδας εργασίας ε, της UEIUNL. Και επίσης τον κύριο Αμαντού Κανούτε, ο οποίος είναι ε, εκτελεστικός ε, διευθυντής του ΣΥΚΟΤΕΒ Αφρικα για την ε, ανάπτυξη και τη συνεργασία. Δίνω το λόγο στον κύριο Διντιέ Νουρισά για 10 λεπτά. Πρόεδρε και συντονίστρια. Σας ε, χαιρετίζω καταρχήν και μας τιμά ιδιαίτερα το ότι μας δεχόσαστε εδώ μέσα στα πλαίσια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Συμβολεογράφων. Γιατί ο συμβολεογραφικός κλάδος ενδιαφέρεται για αυτό το ζήτημα για τις αναπτυσσόμενες χώρες ως προς το καθιστός εγγύου ιδιοκτησίας, διότι διενεργούνται έρευνες και μελέτες σε παγκόσμιο επίπεδο, στην Ευρώπη, Αφρική, Ασία και αλλού. Τα συστήματα χρήσης, ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκές χώρες, μας οδηγούν σε μία περίπου απόλυτα ασφάλεια γιατί στην Ευρώπη έχουμε ένα απόλυτα ασφαλές σύστημα. Διότι τα το σύστημά μας βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας ορίζει το αγαθό. Υπάρχει κτηματολόγιο, υπάρχουν αεροφωτογραφίες, οι φωτογραφίες από δορυφόρους. Το, ο δεύτερος πυλώνας είναι ο νομικός σύνδεσμος που ορίζεται μεταξύ τη γη και το φυσικό πρόσωπο μέσω βεβαίως και της δουλείας και των δουλειών που υπάρχουν και τη μεταβίβαση τίτλων. Ο τρίτος πυλώνας είναι τα δημόσια μητρώα και εκτιματολόγια που συλλέγουν πληροφορίες για τα αγαθά και τα πρόσωπα. Και το σύστημα αυτό είναι αρκετά αποδοτικό για τους εξής λόγους. Γιατί υπάρχει νομική ασφάλεια και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αποδείξουμε ότι το χι αγαθό ανήκει, ανήκει στο ψι ε, φυσικό πρόσωπο, τη στιγμή που κάποιος είναι ιδιοκτήτης της μπορεί να εγγυηθεί με βάση αυτό το αγαθό και να προβεί σε δανειοδοτήσεις ή σε δανειοληψίες και τα κράτη μπορούν να ορίσουν και το φορολογικό καθεστώς για τη συμμετοχή αυτή. Άρα αυτός είναι ο πυρήνας της εργασίας μας. Δεν θέλουμε να εξάγουμε ή να εξαγάγουμε το σύστημά μας, απλώς οι υποανάπτυξη χώρες να το χρησιμοποιήσουν, εάν το επιθυμούν, χρησιμοποιώντας αυτούς τους τρεις πυλώνες διασφάλισης. Όταν αγοράζουμε ένα σπίτι ή γη στις υποανάπτυξη χώρες, δεν υπάρχει αυτή η διασφάλιση, όπως είπε και η Εύα Ζολή. Έχουμε διενεργήσει πολλές ακροάσεις στο Τόγκο, στη Μαδαγασκάρη, στην Τινησία και στην Αϊτή και είδαμε ότι πόρο απέχουμε από αυτή την εξασφάλιση. Ο πρώτος λόγος έγκυται στο εξής. Στην Αφρική το 20% των γεών ορίζονται από κτηματολόγιο, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει διασφάλιση των γεών. Ξέρουμε ότι το 60% των διαφορών στα δικαστήρια είναι, αφορούν την έγκυο ιδιοκτησία. Δεύτερον, υπάρχει το κτηματολόγιο εγκύου ιδιοκτησίας που όρισαν οι άπικοι, αλλά το οποίο δεν προσαρμόζεται στην πραγματικότητα των ελόγω χωρών. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε την κατάσταση των γεών όπως εξελίσσεται. Όταν επινοήθηκε αυτό το σύστημα ήταν εύκολο ένας έπικος ή άπικος να ορίσει 3.000 εκτάρια και να πει ότι είναι δικά του. Αλλά όταν μιλάμε για επιμερισμό εκταρίων, το ζήτημα περιπλέκεται. Ως προς τους ε, τίτλους και την τιτλοποίηση, πρόκειται για 300 με 600 ευρώ που θα πρέπει να καταβάλει κάθε ενδιαφερόμενος και μέσα σε 6 μήνες έως 6 χρόνια μπορεί κανείς να φέρει τον τίτλο αυτό. Χρειάζονται 6 διαδικασίες στο Τόγκο, 23 ε, στη Μαδαγασκάρη και ούτω καθεξής. Έχουμε να κάνουμε με μία ε, δύσκολη και διεφθαρμένη κυβέρνηση ή διακυβέρνηση και υπάρχουν επιμέρους ε, διακυβευόμενα συμφέροντα. Υπήρχαν και ψευδείς τίτλοι που είχαν ε, κατανεμηθεί μέσα στο πλαίσιο αυτό. Επίσης, δεν λαμβάνουμε υπόψη μία νομική πραγματικότητα και χορηγούνται τίτλοι που δεν είναι διασφαλισμένοι ή εξασφαλισμένοι. Επίσης υπάρχουν εναλλακτικά συστήματα τιτλοποίησης για την εξασφάλιση της εγγύου ιδιοκτησίας και αυτό το βλέπουμε στα γκισέ εγγύου ιδιοκτησίας της Μαδαγασκάρης. Ο φίλος μου Αρισού θα σας τα αναλύσει. Ο τρίτος πυλώνας αφορά το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται στο σύστημα εγγύου ιδιοκτησίας που διέπει μια χώρα. Και όπως είπε και η πρόεδρος και η συντονίστρια, θα πρέπει να υπάρχει εξασφάλιση τίτλων, ε, οι οποίοι αφορούν 5-6 στάδια και ούτω καθεξής. Και μόταν όταν υπάρχει ασφαλής τιτλοποίηση δεν υπάρχουν και κλειδονισμοί. Αυτό έχει σχέση και με τα δικαιώματα των γυναικών, διότι στον αγροτικό κόσμο οι γυναίκες είναι επικεφαλής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και χωρίς ε, τίτλους δυστυχώς μπορούν να εκδιωχθούν. Αν διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας, κανείς δεν μπορεί να τις εκδιώξει. Επίσης, οι πλέον ευάλωτοι μπορούν να αποδείξουν τα δικαιώματά τους σε σχέση με επιχειρήσεις ή πλούσιους φορείς που επιθυμούν, να, επιθυμούν την απομάκρυνσή τους. Άρα πιστεύω ότι είναι καλύτερα να υπάρχει τίτλος και όχι δικαίωμα χρήσης ή επικαρπίας. Έτσι μπορούμε να καταπολεμήσουμε την υπεξαίρεση γεών, στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Εύαζολη που γίνεται από ξένες επιχειρήσεις. Και έτσι μπορούμε να ρυθμίσουμε τις συμβάσεις εκμετάλλευσης ή γεωχρησίας. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε σωστή συμβατική πλαισίωση που θα είναι θωράκιση κατά της υπεξαίρεσης και εμπορίας γεών. Εάν το δικαίωμα στη γη είναι κάτι πολύ σημαντικό για τις υποανάπτυξη χώρες, θα δούμε στη συνέχεια ότι και το δικαίωμα στέγης θα αποτελέσει πρόβλημα, ιδιαίτερα στην Αφρικανική Ήπειρο. Ξέρετε ότι στην Αφρική ο πληθυσμός που ήταν της ε, τάξης των 90 ε, των 900 εκατομμυρίων είναι της τάξης του 1 δις, δις 200 εκατομμυρίων στη συνέχεια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αγροτικές εκτάσεις είναι πολύ μεγάλες σε σχέση με τα αστικά κέντρα. Και αν δεν θέλουμε να υπάρξει ένα πολιτιστικό ε, σοκ και ένα σοκ μεταφοράς γεών θα πρέπει να υπάρχει τιτλοποίηση. Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεισφέρει στον τομέα εγγύου ιδιοκτησίας. Μπορούμε να προβάλλουμε μεταρρυθμίσεις με ορισμένες ε, βασικές αρχές. Πρέπει να ενθαρρύνουμε προγράμματα όπου υπάρχει απόλυτη συνεργασία των ρυθμιστών εγγύου ιδιοκτησίας, δηλαδή από πλευράς και οικονομίας αλλά και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Θα πρέπει ανθρωπολόγοι, ε, κοινωνιολόγοι, τοπογράφοι, άνθρωποι της δικαιοσύνης, συμβολεογράφοι να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία δεν θα πρέπει να υπάρχει τομεακός ε, διαχωρισμός. Σε μία χώρα τι κάνουμε, αλλάζουμε το κτηματολόγιο, αλλού το νόμο, σε μία τρίτη χώρα την δημόσια διοίκηση, αλλά αυτό δεν αρκεί. Χρειάζεται ένα ευρύτερο σχέδιο. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι οι συμβολεογράφοι είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουν και επίσης, ευρωβουλευτές θα ήταν σκόπιμο να επισκεφθούν αυτά τα αγγισέ εγγύου ιδιοκτησία στη Μαδαγασκάρη για να δουν πώς υπάρχουν εναλλακτικέ μέθοδοι διασφάλισης των τίτλων εγγύου ιδιοκτησία. Σας ευχαριστώ πολύ. Pardon. <laughs> Donc, euh, merci beaucoup. Ευχαριστούμε πολύ. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Νουρισά, που είναι ο αντιπρόεδρος της ομάδας εργασίας για την τιτλοποίηση της Διεθνούς Ένωσης Συμβολεογράφων. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρα. Είμαι ο Αμπτουλαϊέ Γαρισού, ε, είναι πρόεδρος ομάδας εργασίας τιτλοποίησης ε, των, ε, του Διεθνούς, της Διεθνούς Ένωσης Συμβολεογράφων. Ε, οι προλαλήσαντες ε, εξήγησαν το πρόβλημα. Το πρόβλημα στην Αφρική είναι ότι πριν από την ε, απεικιοκρατία υπήρχε το εθνικό δίκαιο, ήταν συλλογική γη, ήταν ιερή και ήταν στη διάθεση των ανθρώπων για να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν, να την καλλιεργήσουν για να φάνε. Επομένως δεν μπορούσε σε έναν άνθρωπο να ανήκει το Ισλάμ στην αρχή, μετά η δυτική απεικιοκρατία ε, ουσιαστικά αποκριστάλλωσαν τις ε, θεωρίες αυτές. Ε, υπάρχουν όμως ε, παράλληλα με τον, με τον τίτλο έγκυας ιδιοκτησίας, δηλαδή υπάρχει ένα, ε, ένα βιβλίο εγγύου διοκτησίας ε, ε, που είναι κατάλοιπο της Αυστραλίας και είναι ουσιαστικά ισχύει παράλληλα μαζί με το εθνικό δίκαιο και το σύγχρονο δίκαιο το οποίο κληροδοτήθηκε από την απεικιοκρατία πολλοί ανθρωπολόγοι, πολλοί εθνολόγοι θέλουν να παραμείνουμε σε αυτό το εθνικό δίκαιο. Το γνωρίζω αυτό, όμως δεν είναι δυνατόν σήμερα να παραμείνουμε σε αυτό το εθνικό δίκαιο, γιατί υπάρχει καταρχάς ε, η διαφορά των πολιτισμών ε, γιατί υπάρχουν 280, 280 εθνότητες στο Καμερούν σήμερα. Αυτό σημαίνει 280 εθνικά δίκαια. Το ένα αντιμάχεται το άλλο. Τι συμβαίνει. Σήμερα ήρθαν τα χρήματα να διαφθείρουν τις παραδόσεις ε, ε, ε, στο παρελθόν. Ο λόγος ήταν, ήταν νόμος. Σήμερα όμως υπάρχει από τους παραδοσιακούς ηγέτες μία εκμετάλλευση του θυμικού δικαίου και αυτό είναι ένας λόγος ανισότητας. Η γυναίκα επίσης δεν έχει δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Το 2012 δηλαδή δεν μπορούμε να δεχθούμε κάτι τέτοιο είναι επίση όλα προφορικά. Και αυτό είναι πρόβλημα. Και γι' αυτό δεν πρέπει η Αφρική να παραμείνει στο εθνικό δίκαιο. Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα, το σύστημα του ε, τίτλου γης, ε, το οποίο έχει δείξει τα όρια του. Βλέπουμε σήμερα ότι η πρόσβαση των ε, μειονεκτούντων πληθυσμών ε, είναι ελάχιστη. Υπάρχουν ε, τεράστια 95% ε, των καταγγελιών των υποθέσεων που φτάνουν στο δικαστήριο αφορούν αυτό το θέμα. Στο Καμερούν υπάρχουν άνθρωποι που γυρνάνε μετά από τον πόλεμο και βλέπουν ότι άλλοι έχουν πάρει τη γη τους και δεν έχουν κανέναν τρόπο να αποδείξουν ότι αυτή γη είναι δική τους. Και ο μόνος τρόπος που έχουν ε, είναι κάποιος, ένας προφορικός λόγος ε, που έχουν και που ε, δεν αποδεικνύει βέβαια τίποτε. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ε, το 95% των, ε, τίτλων, των, της ιδιοκτησίας ε, δεν καλύπτονται από ένα τίτλο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για την Αφρική, γιατί όταν βλέπουμε τον πληθυσμό της Αφρικής που εκθετικά έχει αυξηθεί, αναρωτιέμαι τι θα κάνουμε αύριο, τι θα κάνουν οι νέοι αύριο, όταν βλέπουμε για παράδειγμα τι γίνεται ε, με, την, ε, ε, με το ότι καρπώνονται τη γη όχι μόνο οι Ευρωπαίοι και οι Βραζιλιάνοι και οι Κινέζοι. Υπάρχουν, είναι πολλαπλό το πρόβλημα. Υπάρχουν επίσης προβλήματα μεταξύ των κτηνοτρόφων και των γεωργών. Γνωρίζετε ότι στην ακτή ελεφαντοστού το πρόβλημα που δημιουργήθηκε εκεί είναι καταρχάς ένα πρόβλημα γης. Αυτή ήταν η αιτία. Οι γυναίκες δεν έχουν δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Το είπαμε και αυτό. Τι κάνουν λοιπόν οι συμβολιογράφοι. Τι προβλέπουν. Την έγκριση της ε, γης ε, με έναν τρόπο, τη δημιουργία τίτλου της γης ε, με έναν όχι δαπανηρό τρόπο, απλό και ασφαλή. Σήμερα δεν μπορούν οι άνθρωποι να έχουν τίτλο διοκτησίας γιατί είναι πραγματικά ένα τεράστιο αγώνα, όπως είπε ο συνάδελφος Διδιέ. Πώς μπορούμε λοιπόν να έχουμε μία εξασφαλισμένη γη πρέπει να υπάρχει ένα επίσημο έγγραφο που θα δίνουμε στον πληθυσμό με απλό τρόπο σε επίπεδο ε, δήμων. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα όλες οι γεές ανήκουν ε, στο κράτος. Πρέπει να υπάρχει ένα τεκμήριο για μία γη, ιδιοκτησίας για μία γη, ο άνθρωπο που την εκμεταλλεύεται μέχρι αποδείξει του εναντίου να θεωρείται ιδιοκτήτη. Επίση, πρέπει να αποκεντρωθεί σε επίπεδο δήμων, όσο μικρή και αν είναι αυτή η δήμη, την έγκαια ιδιοκτησία. Αυτές οι, οι, οι αυτά τα γκισέ, είναι ε, αυτές που πρέπει να αναλαμβάνουν, όπω στη Μαδαγασκάρη για παράδειγμα, τη διαδικασία αυτή. 1500 τίτλοι ε, πλέον ε, μόνο στη Μαδαγασκάρη ε, δίνονται κεντρικά. Όλοι οι υπόλοιποι δίνονται ε, σε αποκεντρωμένο επίπεδο. Με χαρτογράφηση αέρια, με δορυφορική χαρτογράφηση, με το σύστημα Google για παράδειγμα σήμερα μπορεί κανείς να πάει στον υπολογιστή του και να δει πάρα πολύ, με πάρα πολύ λεπτομέρεια που μένει μπορούμε εύκολα να περιχαράξουμε ε, να περιχαράξουμε μία ε, γη, όμως μπορούμε να το κάνουμε και χωρίς ε, αυτό. Γιατί το να κάνει κανείς ένα κτηματολόγιο, δυστυχώς, και η οριοθέτηση είναι κάτι που στοιχίζει πάρα πολύ. Γι' αυτό πρέπει να αρκεί ένα άτομο να καταθέτει ένα φάκελο σε μια επιτροπή, επιτροπή να διαπιστώνει την ιδιοκτησία του ανθρώπου αυτού για τη γη αυτή, πηγαίνει ε, σε επίπεδο Δήμου μετά το θέμα, ε, μιλάμε για το σχέδιο ε, ιδιοκτησίας, εγγύου ιδιοκτησίας του Δήμου, το τοποθετούμε σε ένα χάρτη, συγκεκριμένα οριοθετούμε τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία και του δίνουμε μία ε, έναν τίτλο. 70 ευρώ στοιχίζει στη Μαδαγασκάρη, ενώ με το σύστημα που έχουμε κληρονομήσει ε, από την, ε, από την περίοδο της απεικιοκρατίας είναι 370 ευρώ και περιμένουμε μέχρι 6 χρόνια για μια χορήγηση ενός τέτοιου τίτλου. Θέλουμε λοιπόν μια καθολική πρόσβαση για, όλη την, το για όλο τον πληθυσμό. Είναι κάτι που θα δοκιμαστεί σε επίπεδο ε, υπαίθρου, αλλά ε, και ε, στις φτωχές γειτονιές των, μεγάλων, ε, των μεγαλοπόλεων της Αφρικής, γιατί έχει οριζόντια αυξηθεί το άστι, αλλά όχι ε, καφέτος όπως γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι διαθέσιμος σε ερωτήσεις για να ε, σας ε, πω περισσότερες λεπτομέρειες αν χρειάζεστε. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Αμαντού Κανούτε, εκτελεστικό σύμβουλο της ΙΚΟΝΤΕΒ Αφρικα. Έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο, κύριε Κανουτέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να σας μιλήσω για την ΣΥΚΟΝΤΕΒ της Αφρικής. Πρόκειται για μια οργάνωση για τον πολίτη, την ανάπτυξη και πρόκειται για μια οργάνωση που βασίζεται στο Ντακάρ, που έχει έδρα το Ντακάρ στη Σενεγάλη για να βοηθήσουμε τους πολίτες να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους, για να ξέρουν τι επιπτώσεις έχει κάθε επιλογή τους σε θέματα κατανάλωσης ε, ως προς το περιβάλλον, την ε, καταπολέμηση της ε, φτώχειας και να ξέρουν κατά πόσο το πρότυπο παραγωγής τους έχει επιπτώσεις στην οικονομία, στην καταπολέμηση της φτώχειας και ούτω καθεξής. Η ΣΥΚΟΝΤΕΒ ε, εργάζεται και συνεργάζεται έτσι ώστε οι πολίτες να είναι συνυπεύθυνοι σε αυτή τη διαδικασία συναπόφαση στην ουσία στη Σενεγάλη μέσα σε 10 χρόνια. 650.000 εκτάρια χορηγήθηκαν σε 17 φυσικά πρόσωπα και 650.000 εκτάρια αποτελούν το 17% των αρρώσιμων γεών. Αν λάβουμε υπόψη όλες τις άλλες απειλές κατά της γης, δηλαδή τις πλημμύρες, τη διάβρωση των παράκτιων περιοχών, την απερίμωση και ούτω καθεξής, καθώς και την ε, την έκρηξη της αστιφιλίας, καθώς και τα υφάλμυρα ύδατα, βλέπετε ότι όλα αυτά έχουν τις επιπτώσεις τους. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για βιώσιμη ανάπτυξη. Μιλάμε για μία πηγή κοινωνικής συνοχής αλλά και κοινωνικής αποδόμησης. Μιλάμε για μία πηγή δημιουργίας φτώχειας και γενικότερης ανασφάλειας. Τα αριθμητικά στοιχεία είναι από το καμίας μελέτης της ΣΥΚΟΝΤΕΦ το 2010. Τι έλεγε αυτή η μελέτη. Ότι οι πληθυσμοί που αποχώρησαν από τις γέες τους βρέθηκαν σε μια κατάσταση διατροφικής ανασφάλειας και μία ανασφάλεια για τις ε, γυναίκες που δεν έχουν πια πρόσβαση στη ε, βιομάζα που παρήγαν ε, τα δάση. Και μην ξεχνάμε ότι το 80% αυτής της βιομάζας χρησιμοποιείται για ενεργειακές ανάγκες. Δεν υπάρχει λοιπόν ούτε συγκομιδή, σωστή ούτε σωστή καλλιέργεια γεών. Γι' αυτό η ΣΥΚΟΤΕΒ ζήτησε να σταματήσει αυτή η φαρπαγή υγεών και να γίνει μια σωστή διαβούλευση για να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να υπάρξει μια μεταρρύθμιση εγγύου ιδιοκτησίας και καθεστώτος που διέπει την έγκυο ιδιοκτησία. Να αλλάξουμε λοιπόν το όραμά μας, όπως ισχύει για τα εδαφικά, τα χωροταξικά και ούτω καθεξής. θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις πέντε λειτουργίες της γης. Η γη τρέφει τους ανθρώπους, δημιουργεί απασχόληση, προστατεύει τους φυσικούς πόρους, δημιουργεί πόρους για το κράτος και δημιουργεί πλούτο για τους επενδυτές. Κρίνουμε ότι δεν θα ήταν κατάλληλο να υποσκελίσουμε άλλους τομείς υπέρ του ενός χωρίς να γίνουν διαβουλεύσεις με βάση την επιλογή μας. Δηλαδή δεν πρέπει να επικρατήσει, να δεσπόζει μία επιλογή έναντι των άλλων τεσσάρων. Από αυτόν τον ε, πολυσχηματικό χαρακτήρα και πολυσχηδή χαρακτήρα λειτουργίας της γης, βλέπουμε ότι το 64 υπήρχε μια σύνεση που διείπε αυτό το καθεστώς. Δηλαδή η γη πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό που να ανήκει σε όλους. Η γη ανήκει στο έθνος και το κράτος είναι ο κάτοχος αυτού του δικαίου, αλλά δεν είναι ο απόλυτος, ο απόλυτος συγγνώμη, δεσπότης Άρα βασιζόμαστε στην δωρεάν πρόσβαση στη γη, στη στο, στην ε, έλλειψη ιδιοκτησιακού καθεστώτος, στο ότι δεν μπορεί κανείς να πει σε ποιον ανήκει και σε ποιον μεταφέρεται η γη και οι τοπικές συλλογικές οργανώσεις ορίζουν το ιδιοκτησιακό συλλογικό καθεστώς ελέγχθη με βάση τον πρόσφατο νόμο ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση της εγγύου ιδιοκτησίας. Ανακοινώθηκε και προβλέφθηκε για το 2006, αλλά μέχρι σήμερα δεν είδε το φως της ημέρας. Δημιούργονται όμως άλλα διακυβεύματα. Η παλαιά κυβέρνηση η παρελθούσα κυβέρνηση μέχρι το 2000, από το 2000 μέχρι το 2010 δημιούργησε τις μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις με απελευθέρωση του γεωργικού τομέα και της αγοράς. Άρα η θέση του αγρότη είναι προσβάσιμη στα μεγάλα κεφάλαια που έχουν τη δυνατότητα εκμετάλλευσης. Άρα το 70% των αγροτών δεν μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ μιλάμε για γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Δεύτερον, η μεταρρύθμιση εγγύου ιδιοκτησίας που θα έπρεπε να ισχύει από το 2006 δεν εφαρμόστηκε. Δεν συντάχθηκε καν. Και βλέπουμε ότι 650.000 εκτάσεις δόθηκαν σε 17 φυσικά πρόσωπα της αλοδαπής. Άρα θα πρέπει να σταματήσει αυτή η κατανομή της γης κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλιώς τι θα συμβεί. Όταν θα ισχύσει η μεταρρύθμιση δεν θα υπάρχουν πλέον γης προς κατανομή, γιατί θα έχουν αποδοθεί στους μεγάλους εκμεταλλευτές γης. Το αίτημά μας είναι βάσιμο, γιατί οι συλλογική τοπικοί φορείς δεν έχουν τέτοιες δυνατότητες και αυτό το έχουμε προαναφέρει. Δηλαδή βρίσκονται στο έλεος των πολιτικών δυνάμεων. Άρα χρειαζόμαστε ένα πρότυπο που να λαμβάνει υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία. Το τελευταίο στοιχείο ποιο είναι τα κράτη μας υφίστανται μεγάλες πιέσεις από εταίρους και διεθνείς οργανισμούς που θέλουν την ιδιωτική διαχείριση των γεών. Ποια είναι η επιλογή μας λοιπόν. Η επιλογή μας είναι να εξασφαλίσουμε τις γεωργικές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Και όταν συζητούμε με τους επικεφαλείς των ατομικών εκμεταλλεύσεων μας λένε τι. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε τις υγιές μας, να υπάρχει δικαίωμα χρήσης με βάση το προγονικό δίκαιο, αλλά δεν έχουμε ένα έγγραφο που να, μας, που να αποδεικνύει ότι μας ανήκουν αυτές οι υγιές. Πέρα όμως από αυτό, μας λένε ότι ζουν σε μια κατάσταση επισφάλειας και μέσα στη φτώχεια. Άρα όταν μας ανήκουν αυτές οι γές, όταν έχουμε ιδιοκτησιακούς τίτλους, θα μπορούμε σε περίπτωση ευαλωτότητας να μπορέσουμε να μεταπολίσουμε αυτές τις γές. κάτι το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα. Άρα χρειαζόμαστε εξασφάλιση και μέσα υπεράσπισης και διασφάλισης ιδιοκτησίας. Και γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από τα κράτη να δεχτούν το πρωτόκολλο του Μαπούτο, δηλαδή το 10% του εθνικού προϋπολογισμού να διατίθεται για την αγροτική εξασφάλιση, για την αγροτική πολιτική και ιδιαίτερα για τους ε, μικρούς γεωκτήμονες. Έτσι ώστε να φύγουν από αυτή την επισφάλεια που τους διακατέχει, να έχουν έναν τίτλο ιδιοκτησίας που δεν έχουν αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους που θέλουν βεβαίως να σχολιάσουν. Non. Monsieur Cortés. Κύριε Κορτές. Ευχαριστώ καταρχήν. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω όλους τους ε, πάνελιστ, να τους καλωσορίσω και να σας πω, να τους πω ότι μας ε, ε, διαφώτισαν για αρκετά ζητήματα. Έχω τρεις ερωτήσεις. Ως προς την προσπόρηση που έρχεται από τη γη, την απόδοση της γη. Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο αυτή η μέθοδος δεν είναι πολύ αναπτυγμένη, ιδιαίτερα αναπτυγμένη. Πώς ορίζεται η απόδοση της γης από το κράτος ή από τους ιδιοκτήτες, τους μεγαλογεοκτήμονες. Θα ήθελα να πω στον κύριο, στον κύριο Κανουτέ ότι Κατανοώ ότι υπάρχει πίεση από τα κράτη Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ανταλλαγή γεών, να δούμε ποια θα είναι η σωστή χρήση της γης. Δεν θα θέλαμε η, μας, η αναπτυξιακή μας βοήθεια να σχετίζεται με τις πιέσεις αυτές για την ε, υπεξαίρεση ή κακή χρήση γεών. Και θα ήθελα να ζητήσω τον ε, επικεφαλής των συμβολεογράφων ε, να τον ρωτήσω, υπάρχει κάτι που διέπει το ευρωπαϊκό δίκαιο και που θα μπορούσε να ισχύσει. Υπάρχει και το λεγόμενο ουζουκάπιο, δηλαδή η χρησικτησία. Υπάρχουν ε, αγρότες που εργάζονται για 20 χρόνια πάνω στη γη και θεωρούνται χρησικτήτες χωρίς αυτό να έχει ιχνηλατηθεί από το κράτος. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω κατά πόσο θα μπορούσαμε να προωθήσουμε και αυτή την πτυχή του θέματος, δηλαδή αυτή που στην ουσία εργάζονται πάνω στη γη, κατά πόσο μπορούν να θεωρηθούν χρησικτήτες μετά από 20 χρόνια. Χρόνια, Bergman. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω ε, κι εγώ. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό που είπε ο συνάδελφος από τη Σενεγάλη, επειδή γνωρίζω αυτή τη χώρα λιγάκι. Δύο ερωτήσεις. Πρώτον, η Oxfam ζήτησε μία αναστολή ε, της, ε, των επενδύσεων στις ε, ε, γέες ε, από τις ε, ε, πολυεθνικές, από τις διεθνείς εταιρείες. Επίσης, ποια είναι η άποψή σας όσον αφορά την έλλειψη του δικαιώματος των ντόπιων γεωργών λόγω της αναγκαιότητας βελτίωσης του δικαιώματος ιδιοκτησίας των γεών. Μιλήσατε και για το κτηματολόγιο. Είναι άποψή σας λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ε, ότι ε, μπορεί ε, στο πλαίσιο των δράσεων που είναι δυνατόν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Κατσμάρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για τις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις τους. Έχω μία ερώτηση και μία παρατήρηση. Καταρχάς μία ερώτηση προς τον τελευταίο ομιλητή, τον κύριο Κανούτε αυτό το αίτημα για 10% επενδύσεις στον αγροτικό τομέα δεν είναι τίποτα καινούριο. Η Ένωση Αφρικανικών Χωρών το έχει επαναλάβει αυτό πολλές φορές και έχει κάνει έκκληση ε, με την οποία συμφωνώ απολύτως στις κυβερνήσεις των μελών χωρών. Ρωτώ όμως, γιατί αυτό συνεχίζει να συμβαίνει. Ξέρουμε τόσα χρόνια ότι έχουμε, έχει υποβληθεί αυτό το αίτημα, ε, το επίγον αίτημα στις κυβερνήσεις και τίποτα δεν έχει γίνει. Επίσης, ότι όσον αφορά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των ε, μικρών παραγωγών, των μικρών ιδιοκτητών, εγώ προέρχομαι από ένα κράτος όπου πρόσφατα υλοποιήθηκε μία αγροτική μεταρρύθμιση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτή η αγροτική μεταρρύθμιση συμπεριέλαβε δύο πολύ σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, ε, βασίστηκε στην πολιτική βούληση, διότι αν υπάρχει πολιτική βούληση ε, μπορεί να ακούσει ε, τη φωνή της βάσης, δηλαδή τη φωνή του, του, του λαού. Ε, ο λαός πρέπει να πιέσει για να δημιουργηθεί πολιτική βούληση για μεταρρύθμιση. Και επίσης βασίστηκε στην τακτοποίηση της τεκμηρίωσης δεν μπορεί βεβαίω ευθύ εξ αρχή να βρεθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, αλλά σιγά σιγά θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα καθεστώ που να αποδεικνύει ότι υπάρχουν αυτά τα χαρτιά που αποδεικνύουν την ιδιοκτησία. Επαναλαμβα... Επανέρχομαι λοιπόν στο πρώτο μου ερώτημα. Υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση που προέρχεται από την πίεση της βάσης του πληθυσμού, της βάσης των ιδιοκτητών, των παραγωγών, ε, των, μικρο, των μικροεκμεταλλεύσεων. Υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση. Η λύση βρίσκεται, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν λύσεις αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Μάλιστα. Ήδη υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Καλύτερα να δοθούν τώρα οι απαντήσεις. Δεν ξέρω ποιος θέλει να απαντήσει πρώτος. Κύριε, Αρισού, κύριε Νουρίσα, ε, ε, ευχαριστώ πολύ. Στη σχέση τώρα με την, ε, το μορατόριουμ για την αρπαγή των γεών, θα ήθελα να πω το εξής. Δεν μπορούμε να φανταστούμε μία ξένη εταιρεία σε μία ξένη χώρα να αρπάζει γη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια συμβατική σχέση μεταξύ των χωρών και των εταιριών. Τότε μπορούμε να πλαισιώσουμε, να ρυθμίσουμε και να ελέγξουμε. Καλό είναι το μορατόριο, αλλά δεν νομίζω ότι στην πράξη ε, περιγράφει πολύ καλά τι θέλουμε να κάνουμε. Αυτό που είπε ο κύριος Κατσμάρεκ, η πολιτική βούληση προσκρούμε σε κάθε προσπάθειά μας, σε μια έλλειψη ε, βούλησης από τις χώρες. Για παράδειγμα, δρομολογήσαμε ένα πρόγραμμα ε, να συνοδεύσουμε στην ΑΕΤ ένα, ένα, ένα πρόγραμμα ε, ε αρπαγής, ε, κατά της αρπαγής των γεών μετά το φοβερό σεισμό του 2010 ε, κάναμε μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά ε, για το ζήτημα της, ε, των γεών και τελικά άλλαξαν όλα γιατί άλλαξε ο Πρωθυπουργό και θέλει να πάρει, να καρποθεί όλα τα κονδύλια που είχαν προβλεφθεί. Είναι κρίμα αξιοθρύνητο και μας χαλάει εντελώς ε, και κάθε προσπάθεια. Εδώ και τέσσερις, ε, τέσσερα χρόνια κάνουμε lobbying ε, και στην κυβέρνηση και στους βουλευτές για να υπάρξει μια πραγματική ε, μια δέσμευση πραγματικής αναθεώρησης ε, της, ε, του καθεστώτος, του εγγύου καθεστώτος, μόνο όμως αν τους πείσουμε ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, πραγματικά κάθε φορά προσκρούμε σε έναν τοίχο. Και ένα τελευταίο που θα θέλαμε να πούμε, ο συνάδελφος Αρισού θα συμπληρώσει άλλωστε και αυτά που λέω, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως τώρα. Όταν πηγαίνουμε στις ε, ξένες ε, χώρες ε, και ξέρουμε ότι έχουμε μεταβεί σε πολλές χώρες, Μαδαγασκάρι, Μπουρκίνα Φάσο, Τόγκο, Αϊτή κλπ. Κάθε φορά επισκεπτόμαστε τους εκπροσώπους επιτόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως σε γενικές γραμμές το θέμα της εγγύου ιδιοκτησίας δεν τους απασχολεί πάρα πολύ και είναι κρίμα, γιατί είναι σημαντικό τμήμα της οικονομικής ανάπτυξης των χωρών αυτών. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Κύριε Αρισού, ευχαριστώ πολύ. Για να απαντήσω στο δεύτερο τμήμα της ερώτησης του ε, κυρίου Κορτές για το δικαίωμα ε, ενοικίασης γης. Υπάρχει κάποιο είδους ε, σύστημα στην Ιγυρία αν, αν κάποιος θέλει να χτίσει ένα σπίτι κάπου 90 χρόνια είναι το δικαίωμα ιδιοκτησίας. Τώρα για εμπορική εκμετάλλευση, ε, όπως για παράδειγμα ένα βενζινάδικο, είναι 40 χρόνια. Είναι όμως ε, ε, ένα συμβόλαιο σαν ε, όλα τα υπόλοιπα και ο ιδιοκτήτης είναι το κράτος και με τη διαφορά Έξι μήνες έχει κανείς, για παράδειγμα, στη διάθεσή του για ανανέωση. Αν δεν το ζητήσει σε πέντε μήνες, 29 ημέρες, χάνετε την ιδιοκτησία σας. Όμως υπάρχει το εθιμικό δίκαιο, οι εθιμικοί κανόνες, οι οποίοι αναγνωρίζονται μεν, όμως πρέπει να περάσει κανείς μέσα από αυτό το, δικαιό, το, το, το εθνικό δίκαιο σε ε, αυτό το, ε, αυτή την ιδιοκτησία της γης, ενός είδους συμβόλαιο τέλος πάντων, ε, για 90 χρόνια όμως ε, τα εδάφη, τα βοσκοτόπια για παράδειγμα, από 12 χιλιόμετρα από την πόλη δεν έχει καν δικαίωμα σε συμβόλαιο κανείς. Οπότε σιγά σιγά εξαφανίζονται οι, τα βοσκοτόπια και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους ε, κτηνοτρόφους και τους ε, γεωργούς στις ε, αγγλόφωνες χώρες, στις γαλλόφωνες χώρες. Αυτού του είδους το σύστημα ισχύει μόνο σε περίπτωση ε, εκβιομηχάνησης ε, γιατί ε, δίδεται η γη στους διάφορους ιδιοκτήτες ανάλογα με την περίπτωση. Ε, και αυτό το θέμα περνάει από τον Πρωθυπουργό, μετά από έναν Υπουργό κλπ. Και έτσι ενισχύεται η αρπαγή της γης. Δεν υπάρχει δικαίωμα ε, ε, κυριότητας της γης για την εκμετάλλευση, τουλάχιστον στις γαλλόφωνες χώρες, ούτε στις Σενεγάλη. Όσον αφορά τώρα το θέμα που έθεσε ο δεύτερος βουλευτής που μίλησε για το μορατόριουμ της Oxfam, κοιτάξτε, αυτό που ζητήθηκε είναι τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω, λοιπόν, να, κάνουμε, να το θεωρήσουμε μία προϋπόθεση αναπτυξιακής ε, βοήθειας όπως έχουμε ρήτρε ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, κλπ. Να υπάρχει και αυτή η ρήτρα μία χώρα που ζητά βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να δεχθεί αυτή την απαραίτητη προϋπόθεση, διαφορετικά δεν υπάρχει το δικαίωμα στη βοήθεια. Αυτό είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα οι πληθυσμοί δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Ο κύριος Κανούτε το είπε. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κανούτε είναι η αιτία της, ε, του προβλήματος στην Αφρική. Το Τόγκο, η Σενεγάλη και το Καμερούν ε, ενέκριναν τον ε, δημόσιο τομέα. Όμως πρέπει να δείξει κανείς πρώτα ότι πριν από το 1974, όταν άρχισε να ισχύει το συγκεκριμένο κείμενο, είχε κανείς αυτή τη γη στην ιδιοκτησία του. Ε, είναι όμως πολύ δαπανηρό το σύστημα, υπάρχει και η διαφθορά και σήμερα αυτό που συμβαίνει είναι ότι 90% των γεών δεν είναι αντικείμενο τίτλου γιατί όταν κάποιο, ας πούμε, βγάζει ένα δολάριο, ένα ευρώ την ημέρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο 400 ευρώ να εξοδεύσει. Δηλαδή, ολόκληρο το, ε, ε, το εισόδημά του για ένα χρόνο για να αποκτήσει έναν τίτλο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ούτε έχει το χρόνο να περάσει από όλη αυτή τη μακροχρόνια διαδικασία. Θέλει να πάρει ε, λίπασμα, να πάρει ε, ε, κάτι άλλο που χρειάζεται για την ε, καλλιέργεια. Όχι όμω να ξοδέψει αυτά τα χρήματα για να πάρει έναν τίτλο. Υπάρχει ένα πρόβλημα πολιτική βούληση και το λέω αυτό γιατί μιλάμε σήμερα, συνομιλούμε συνεχώ με του ε, γαλλόφωνου εταίρου μα στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού ε, ε, Γαλλοφώνων και στο Κοτονού είχαμε μία συμφωνία που προβλέπει ότι θα υπάρξει μία επιτροπή που θα έχει το καθήκον ε, σύνταξης ενός κειμένου 15 άνθρωποι που θα προέρχονται από τον τομέα το συμβολεογραφικό, ε, και άλλοι εμπειρογνώμονες, ε, ε, νομομαθείς της Κεντρικής και Δυτικής Αφρικής, με 8 τεχνικούς, με τοπογράφους, έναν Ευρωπαίο, έναν Αφρικανό, με κοινωνιολόγους, με ανθρώπους της πληροφορικής, της χαρτογράφησης κλπ. για να υπάρξει ένας νόμος πλαίσιο που θα ισχύει για όλες τις γαλλόφωνες χώρες τουλάχιστον σε μία πρώτη φάση μετά μπορεί να εγκριθεί και να ισχύσει και στις υπόλοιπες χώρες. Αυτό το νόμο πλαίσιο το χρειαζόμαστε υπερεθνικό. Ξέρετε ότι σήμερα ε, το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε στην Αφρική ε, ή και άλλα δικαιώματα είναι τμήμα ε, ενός συγκεκριμένου οργανισμού που ασχολείται με τα δικαιώματα αυτά αυτό επιτρέπει να υπάρχει μια ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ε, ε, κείμενα δηλαδή που είναι πέρα από την εθνική επιρροή. Κάτι τέτοιο θα δώσει τη δυνατότητα στους επενδυτές να εξασφαλίζουν όχι απολύτως, αλλά τέλος πάντων με πιο αποτελεσματικό τρόπο τις συναλλαγές τους ε, στην Αφρική. Αυτή την πολιτική βούληση λοιπόν εμείς τη χρειαζόμαστε και τη ζητούμε μέσω των ε, βουλευτών. Ο κύριος Κατσμάρικ έχει δίκιο όμως. Χρειάζεται οπωσδήποτε πολιτική βούληση και εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν συμπεριλάβει μια τέτοιου είδους ρήτρα ε, στη βοήθεια την αναπτυξιακή, μπορεί να πιέσει τις αφρικανικές κυβερνήσεις, ε, γιατί ε, πάντοτε η κυβέρνηση στέλνει τα σχέδια νόμου, ουσιαστικά απλώς καταγράφουν τα κοινοβούλια στις αφρικανικές χώρες. Εμείς χαιρόμαστε που οι Αφρικανοί βουλευτές υποστηρίζουν την ιδέα αυτή, αλλά δεν είναι δεδομένο ότι αν δεν τις υποστηρίξουμε μέσω οργανισμών όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα καταλήξουν κάπου αυτές οι προσπάθειες. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Για δέκα δευτερόλεπτα σας δίνω το λόγο. Κύριε Χαρισού, Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας, γιατί είναι διαβιέστατες. Αλλά το να αμφισβητεί κανείς την αναπτυξιακή βοήθεια δεν είναι και κάτι τόσο δημοφιλές. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση η, ευκολία με την οποία θίγεται το θέμα. Ο κύριος Κανούτε. Το moratorium... ορίζει αυτό που εμείς είχαμε ζητήσει εδώ και τρία χρόνια. Τασόμαστε υπέρ αυτού του μορατόριου. Θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή άμεσα, έτσι ώστε τα κράτη να κινηθούν προς την μεταρρύθμιση αυτή, συνενετικά. Δεν μπορούμε με βάση τις πέντε λειτουργίες της γης απλώς να πούμε moratorium, τελεία και παύλα. Δεν μπορούμε να παραχωρούμε τις γιές αλόγιστα. Θα φτάσει μια στιγμή όπου οι άνθρωποι θα πούνε τι γίνεται. Τη στιγμή λοιπόν που χορηγούνται οι υγιές θα πρέπει να υπάρχει διασφάλιση μέσω τίτλων. Γι' αυτό μιλάμε για μορατόριου για να μπορέσουμε τάχιστα να κινηθούμε προς μια συνενετική συζήτηση και να πούμε ότι έτσι βλέπουμε το εδαφικό καθεστώς που πρέπει να μας διέπει. Το 10% θα πρέπει να αφορά τις ε, γές προς κτηνοτροφία, ένα 10% τα ενδιαιτήματα και ούτω καθεξής. Δηλαδή θα πρέπει να δώσουμε μία ποσοστή αναλογία για κάθε λειτουργία. Αυτό το μορατόριο θα πρέπει να έχει μία στοχοθέτηση, κτηματολόγιο. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας. Πρέπει να είμαι προσεκτικός εδώ. Προτιμώ να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε με τις χώρες μας ε, διάφορες πλαισιώσεις συνεργασίες, κοτόνου και άλλες. Και εκεί έχουν ενταχθεί ορισμένες αρχές. Η αρχή της διαφάνειας μας βρίσκει σύμφωνος. Και τα κράτη και την ε, κοινωνία των πολιτών. Άρα στις διαπραγματεύσεις συνεργασίας θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι μηχανισμοί που διασφαλίζουν τη διαφάνεια. Έτσι ώστε να μην υπάρχει διατροφική ανασφάλεια. Να δούμε ποια είναι τα μέσα έτσι ώστε να κατανέμεται η γη με βάση αυτές τις πέντε λειτουργίες. Να μην επιβαρύνει τους μικροαγρότες. Αυτά είναι θέματα αρχής, τα οποία ε, υπερασπιζόμαστε αμφότεροι. Τώρα, η αποκέντρωση μπορεί να γίνει. Μπορούμε με την ησυχία μας να το θέσουμε το ζήτημα. Αλλά ως προς την ερεσιμότητα είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και ευαισθητοποιημένοι. Γιατί το 10% του Μαπούτο δεν ισχύει. Μα είναι θέμα πολιτικής βούλησης, το είπατε κι εσείς. Αλλά είναι και ένα ζήτημα που αφορά <coughs> τις κοινωνικές δυνάμεις που θα συνδράμουν και που δεν ήταν πάντα παρούσες. Υπάρχει σήμερα ένας μηχανισμός εκκίνησης. Η κοινωνία των πολιτών που εκπροσωπεί αυτές τις κοινωνικές δυνάμεις αναλαμβάνει αυτό το έργο. Αυτό είναι το σημείο εκκίνησης, δηλαδή η καταγγελία της υφαρπαγής γεών. Και μέσα στα πλαίσια του δικαιοδοτικού συστήματος, τουλάχιστον σε Σενεγάλη, δεν είναι δυνατόν να ξεχάσουμε τις αγροτικές περιοχές, γιατί μια κυβέρνηση δεν μπορεί να υφαρπάξει τις ε, ΓΕΣ όπως επιθυμεί, χωρίς να υπάρξει αντίδραση της κοινωνίας των πολιτών. Άρα αυτό το 10% εάν δεν, είναι, δεν αποτελεί πραγματικότητα, δεν αποτελεί πραγματικότητα γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Ακόμα και οι χώρες που εφάρμοσαν το 10% θα πρέπει να δούμε κατά πόσο τα, τα σύνολα και οι ομαδοποιήσεις φτάνουν σε αυτό το 10%. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε αν το σύνολο του προϋπολογισμού αντικατοπτρίζει αυτό το 10% και δεν φτάνει σε ένα 4% επί της ουσίας. Ευχαριστούμε πολύ. Τελείωσε αυτό το πάνελ. Ο Έντουαρ Κοζόσνικ έχει το λόγο για το δεύτερο πάνελ. Ευχαριστώ. Ας αλλάξουμε θέμα λοιπόν και γλώσσα. Εκπροσωπώ τους ε, ψηφοφόρους της ε, Τσεχίας και θα διαρωτηθείτε ίσως ε, γιατί προεδρεύω του πάνελ αυτού. Ε, η απάντηση είναι εύκολη. Οφείλεται στο όνομά μου, ε, το οποίο συμπίπτει με το όνομα ε, του, του κυρίου Ντίβα, ο οποίος είναι εμπειρογνώμων, ο μεγάλος εμπειρογνώμων των θεμάτων αυτών, και ο οποίος δυστυχώς, επειδή γίνεται η συνδιάσκεψη του κόμματος των συντηρητικών αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν μπόρεσε να είναι παρόν. Και έτσι ο κύριος Ντίβα ζήτησε να τον αντικαταστήσω εγώ. Τα θέματα αυτού του πάνελ είναι πολύ ενδιαφέροντα και για μένα προσωπικά, διότι προερχόμενος από τη Δημοκρατία της Τσεχίας, ε, περάσαμε κι εμείς μία περίοδο μεταρρύθμισης ε, από τη δεκαετία του 90 και εν ώψη της ε, εντάξεώς μας ε, βεβαίως και γι' αυτό ε, το θέμα του ιδιωτικού τομέα και του ρόλου του στην γεωργία με ενδιαφέρει διακαώς. Έχουμε μεγάλη εμπειρία από τη χώρα μου με τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν και πιστεύω ότι το θέμα του πώς μπορούμε, πώς μπορεί ο ιδιωτικό τομέα να βοηθήσει, να συνδράμει, να συνεργαστεί και να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης της γεωργίας ενδιαφέρει όλους. Δίνω λοιπόν το λόγο στον κύριο Κλέιτον Σέφερ. Είναι η τρίτη φορά που είμαι εδώ και ομιλώ για τα ίδια θέματα, το οποίο κατά κάποιο τρόπο μου δημιουργεί μια στεναχώρια διότι ακούω συνέχεια τα ίδια προβλήματα από τους εκπροσώπους των χωρών αυτών για την ανασφάλεια της εγγύου ιδιοκτησία, για την έλλειψη κτηματολογίου, για το πρόβλημα της κατανομής και διανομής των γεών. Το θέμα είναι λοιπόν πώς θα μπορέσουμε να εδραιώσουμε ένα σωστό κτηματολόγιο, πώς θα μπορέσουμε να καταγράψουμε, να οριοθετήσουμε τις ε, κατά πολύ τεμαχισμένες ιδιοκτησίες, τις ΓΕΕΣ, και πώς θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε συνεχεία τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και να βοηθήσει ένας ε, διεθνής συνασπισμός ενδιαφερομένων να προστατεύσει τους μικρούς παραγωγούς που έχουν τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Είναι λοιπόν το ίδιο πρόβλημα που επανέρχεται συνέχεια στην επικαιρότητα και οι στόχοι μας περαμένουν ήδη. Ακούσαμε πολλά για την Αφρική. Εγώ αυτή τη στιγμή επικεντρώνω τις προσπάθειές μου στην Ινδία. Οι προηγούμενοι ομιλητές του πάνελ εξήγησαν πάρα πολύ καλά τα προβλήματα της Αφρικής, αλλά έχουμε παρόμοια προβλήματα στην Ινδία. Μάλιστα σήμερα 100.000 άνθρωποι διαδηλώνουν στην, στο Νέο Δελχή κατά της υφαρπαγής γεών και των, των μικρών τους χωραφιών δηλαδή που έχουν και καλλιεργούν. Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε ε, μια κατάσταση η οποία είναι καταστροφική για πάρα πολλούς χωρικούς, για πάρα πολλούς μικροκαλλιεργητές. Βεβαίω έχει περάσει ένα στο νομοσχέδιο στην Ινδία πρόσφατα το οποίο διασφαλίζει ε, τη, τα δικαιώματα διοκτησία ε, των ΓΕΑΣ ε, μετά από πέντε χρόνια χρησικτησίας. Μετά από πέντε χρόνια εκμετάλλευσης υπάρχει το δικαίωμα της χρησικτησίας. Όμως 100 εκατομμύρια περίπου μικροπαραγωγή είναι σε αυτή την κατάσταση, οπότε καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται ένα τεράστιο έργο σε με πολλές πτυχές και σε πολλά μέτωπα για να μπορέσει να περάσει περαιτέρω νομοθεσία που να τους διασφαλίζει. Επίσης, ε, αυτή τη στιγμή συζητούμε προγράμματα με την ε, Παγκόσμια Τράπεζα ανάπτυξης ε, της γεωργίας για την παροχή και συνδρομή εμπειρογνωμόνων που θα βοηθήσουν τους μικροπαραγωγούς στο να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Σε αυτό τον τομέα της ε, αγροτικής, ε, τον αγροτικό τομέα, στη γεωργία γενικά, οι ανταγωνιστές είναι συνήθως τεράστιες και παντοδύναμες εταιρείες. Βλέπουμε βεβαίω μια όθηση του αγροτικού τομέα. Από τη μία πλευρά έχουμε τους μεγάλους παίκτες για τα, την παραγωγή τροφίμων, βιοκαύσιμα, για την παραγωγή βασικών ειδών διατροφής κλπ. Στις, στις χώρε. χώρες. Και έτσι βεβαίως καταλαβαίνετε ότι δεν συμφέρει πλέον να είναι κανείς ένας μικρός παραγωγός και υπάρχει ακριβώς αυτή η έξοδος από τις, την Ήπεθρο προς τις μεγάλες πόλεις που τραβάει τους ε, μικροκαλλιεργητές αμαγνήτες. Και γι' αυτό οι μικροκαλλιεργητές, οι μικροπαραγωγοί είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και αντιλαμβάνονται ότι δεν υπάρχουν πιθανότητες να επανέλθουν στις παραδοσιακές ε, ε, καλλιέργειες που είχαν στο παρελθόν ε, όπου παρήγαγαν ε, τα βασικά είδη διατροφής όταν παλαιότερα δίνονταν τεράστιες επιδοτήσεις για αυτές τις καλλιέργειες, για αυτά τα προϊόντα. Πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή να αναγνωρίσουμε ότι γίνεται ένας διαχωρισμός μεταξύ εμπορικής γεωργίας και παραδοσιακής γεωργίας και κάνω μία έκκληση να εξετάσουμε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που ξεκινάει από τον μικρό μεμονωμένο παραδοσιακό παραγωγό μέχρι τον ε, εδρεωμένο μεγάλο παραγωγό στα πλαίσια της βιομηχανικής γεωργίας. Υπάρχουν λοιπόν ε, οργανισμοί που μπορούν να βοηθήσουν τα μέλη τους ε, ε, προγράμματα που βοηθούν τους μικρούς παραγωγούς έτσι ώστε να μπορούν να τους βοηθήσουν μέσα στο τοπικό περιβάλλον στο οποίο κινούνται. Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες, υπάρχουν δυνατότητες ε, διασφάλισης ενός καλού εισοδήματος για τους συμμετέχοντες σε αυτά τα προγράμματα. Δεν είναι απαραίτητο να συνδέσουμε τη χαμηλή παραγωγικότητα με την απελπισία, με την ε, έλλειψη κάθε ελπίδας ε, ευπρεπούς διαβίωσης και, ενός, και εξασφάλισης ενός ευπρεπούς εισοδήματος λόγω του ανταγωνισμού των μεγάλων ε, επιχειρήσεων. Η διασφάλιση των γεών ε, είναι πάρα πολύ, η διασφάλιση της εγγύου διοκτησίας είναι πάρα πολύ σημαντική και η τίτλη βεβαίω για κάποιο παραγωγό, διότι έτσι θα μπορέσει να ξεκινήσει τις αιτήσει του για ε, τα κεφάλαια που χρειάζεται, για τις, ε, την άρδευση, την αγορά των σπόρων και τις πρώτες ύλες. Εάν όμως γνωρίζει ότι η αίτησή του για τη διασφάλιση της εγκύου διοκτησία του, του χωραφιού του δηλαδή και η αίτησή του για την απόκτηση νομίμων τίτλων δεν θα ε, επαληθευθεί, δεν θα εγκριθεί και ότι δεν έχει πιθανότητες, τότε βεβαίως επέρχεται η απεσιοδοξία και η καταστροφή. Επίσης, πρέπει να διασφαλίσουμε την πρόσβαση στις αγορές. Ε, της παραγωγής. Να μπορεί να, να έχει πρόσβαση. Αν δείτε όμως την τρέχουσα κατάσταση είναι σαφές ότι οι μικροί παραγωγοί δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις εμπορικές αγροτικές ε, επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις παραγωγής ε, τροφίμων. Ε, δεν έχουν τη δυνατότητα και τα μέσα. Θα πρέπει λοιπόν οι μικροκαλλιεργητές και οι μικροπαραγωγοί να επικεντρώσουν την προσοχή τους σε, άλλες, ε, σε άλλους τομείς, ε, παραδείγματος χάρη σε διάφορες ε, στη συμπαραγωγή τροφίμων υψηλή ποιότητα ή περιορισμένη ζήτηση αλλά υψηλή διατροφική αξία πρέπει να εξασφαλίσουν ότι μπορούν να συμμετάσχουν σε μία αγορά ε, με ιδιαιτερότητες για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν αλλά αυτό και πάλι θα γίνει μόνο εάν έχουν ασφάλεια ε, της, έγκυου, της και τίτλους. Ακούσαμε κυβερνήσεις που πραγματικά εκδιώχνουν τους ε, παραγωγούς από τις ε, καλλιεργήσιμες γέες, από τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις που είναι και εξαιρετικής ποιότητος συμβαίνει αυτό και πολλές φορές αναγκάζονται οι κάτοικοι που έχουν ένα χωραφάκι ας πούμε αλλά δεν έχουν τους τίτλους να το πουλήσουν σε ένα τρίτο άτομο και συνεχεία να φύγουν θέλουμε η διεθνή κοινότητα να αντιδράσει ενεργά και να σταματήσει αυτό το φαινόμενο του ξεπουλήματος των μικροϊδιοκτησιών σε τρίτους οι οποίοι συνεχεία τα μεταπουλούν αλλά εντάξει φεύγει ο πληθυσμό από την Ήπεθρο διότι αυτό οδηγεί σε εμφύλιους πολέμους. Βεβαίως υπάρχει και η μεγάλη αλλαγή στην αξιολόγηση των αγροτικών προϊόντων, παραδείγματος χάρη τα βιοκαύσιμα Καταλαβαίνετε ότι η καλλιέργεια των βιοκαυσίμων σε τεράστιες εκτάσεις διώχνει τους μικροϊδιοκτήτες ε, των γεών και τους αναγκάζει να γίνουν ε, εργάτες των μεγάλων ιδιοκτητών ε, και καλλιεργητών των νέων προϊόντων. Και, και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση έχουμε ήδη δείγματα ότι οι εξελίξεις θα είναι πάρα πολύ κακές, αρνητικότατες. Τώρα, οι παράγοντες του ιδιωτικού τομέα μπορούν να κάνουν πολλά για να αναπτύξουν αγροτικά συστήματα και να βελτιώσουν την έγκυο ιδιοκτησία, την διτλοποίηση. Η εταιρεία συμβούλων στην οποία εργάζομαι εδώ και πολύ καιρό προτείνει την ε, δημιουργία ενός διεθνού Ινστιτούτου, Διεθνού Ιδρύματος, το οποίο θα μπορεί να παρακολουθεί τα αιτήματα που υποβάλλονται από ανεξάρτητους ε, μικροϊδιοκτήτες και να καταγράφει και αναλύει όλα αυτά τα στοιχεία, μηχανογραφημένα βεβαίως, ε, όλες τις πληροφορίες, ε, έτσι ώστε μέσω των αναπτυξιακών προγραμμάτων να μπορούν να υλοποιηθούν τα προγράμματα ώστε όλα τα στοιχεία αυτά που υποβάλλονται, τα δικαιολογητικά, αν θέλετε, η τεκμηρίωση, να καταγραφούν, να, καταγραφούν, να υπάρχει μια τράπεζα δεδομένων δηλαδή. Που ακόμα και αν δεν υπάρχουν νόμιμοι τίτλοι ιδιοκτησία, τουλάχιστον θα βοηθούν τους ανθρώπους αυτούς στην περαίωση και στη διεκπαιρέωση των φακέλων που έχουν υποβάλει, των ετοιμάτων τους. Επίσης, ε, μπορούμε ενδεχομένως να προσφέρουμε μία ασφάλεια εγγύου ιδιοκτησίας που θα οδηγούσε σε περίπτωση προσφυγής στο δικαστήριο στην καταβολή κάποιας αποζημίωσης σε περίπτωση που ε, χάνει τη γη του. Μην ξεχνάτε ότι οι περισσότεροι μικροκαλλιεργητές ε, δεν έχουν καμία πίστη ε, στη γραφειοκρατία και στις διοικητικές αρχές της χώρας τους, η οποία τους έχει ξεπουλήσει ε, επί χρόνια και δεκαετίες. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη αναξιοπιστία, μεγάλη δυσπιστία από την πλευρά τους. Και αυτή η κατάσταση δεν πρέπει να συνεχιστεί. Αυτά είχα να πω. Ο πρόεδρος του πάνελ. Ευχαριστώ. Ο επόμενος καλεσμένος μας είναι ο κύριος Αλάν Αντίλ, ερευνητής και πρόεδρος του, της Υποσαχάρης Αφρικής του προγράμματος για την Υποσαχάρη Αφρική. Γεια σας, είμαι συντάκτης ε, μιας μελέτης ε, πέρσι για την υποσαχάρη Αφρική. Ε, πραγματικά αφορά 100% το σημερινό θέμα της ακρόασης. Θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα όσον αφορά τον ορισμό και τις συνέπειες των επενδύσεων ε, στις ΓΕΕΣ. Θα ήθελα να σας επιστήσω το προσοχή στο γεγονός ότι όπως ε, είπαμε οι περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε για σύμβασης ε, συμβάσεις εμφύτευσης όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Εγώ θα αναφερθώ μόνο σε ένα τμήμα του θέματος γιατί όταν δούμε τα 200 εκατομμύρια εκταρίων γης που έχουν ανταλλαγή από την αρχή της δεκαετίας του της ε, ε, ε, δεκαετίας του 2000, όπως είπε και η κυρία Ζολή, ένα μεγάλο τμήμα έχει πάει σε ξένους επενδυτές. Εγώ να επικεντρωθώ σε αυτό το σημείο, αλλά δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι το μεγαλύτερο τμήμα των επενδύσεων και των επενδυτών είναι εθνικής φύσεως η θα διαρθρωθεί σε τρία σκέλη ε, η, παρουσίασή μου. Τα δύο πρώτα, το πρώτο μάλλον αφορά τον ορισμό και τη δύσκολη εκτίμηση του φαινομένου, ε, την, ε, την υφαρπαγή των γεών τέλος πάντων, land grabbing, ποιοι είναι οι εταίροι αυτής της επένδυσης. Είναι ενδιαφέρον αυτό γιατί δεν το εξετάσαμε αυτό καθόλου στην ακρόασή μας και θα ολοκληρώσω με ε, τις συνέπειες, ε, πιο μακροσκελές αυτό, ε, των επενδύσεων αυτών. Πρώτον, λοιπόν, η εκτίμηση των επενδύσεων αυτών είναι δύσκολο να έχουμε σωστό νούμερο γιατί το θέμα αυτό ήρθε στο προσκήνιο ουσιαστικά το 2008 λόγω της ε, υπόθεσης στη Μαδαγασκάρη, δηλαδή ότι η εταιρεία η κορεατική μαθαίνει ότι της είχαμε υποσχεθεί ένα εκατομμύριο, μαθαίνουμε ότι της είχαν υποσχεθεί ένα εκατομμύριο εκτάρια, ε, γίνεται κοτζάμ σκάνδαλο, αποσύρεται η εταιρεία, μετά υπήρξε το επισητιστικό θέμα και έτσι ουσιαστικά ε, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή ε, ένα φαινόμενο το οποίο έχει πάρα πολύ επιδεινωθεί και γρήγορα από τις αρχές του 2000. Και επιμένω γιατί οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και εφημερίδες, ε, πολυάριθμες, ε, έθεσαν κάποια δημοσίευσαν κάποια νούμερα τα οποία δεν είναι απολύτως ακριβή. Αν θέλετε αξιόπιστες μελέτες, υπάρχει σίγουρα μια συλλογή ε, κέντρων ε, ε, ερευνητικών με πάρα πολύ αξιόπιστες και αξιέπαινες δημοσιεύσεις, όχι απλώς δηλαδή ανακοινώσεις στις εφημερίδες, δηλαδή 500.000 εκτάρια δόθηκαν σε κάποιον κλπ. κλπ. Είναι πολύ πιο συγκεκριμένα και πολύ πιο πρεσιωμένα για την Ιγυρία, αν προσθέσουμε όλα τα εδάφη για όλα τα προγράμματα, το Δέλτα του Νίγηρα, το Μαλί μιλάμε, 650.000 εκτάρια. 2012 λέει ότι τα ε, προγράμματα ουσιαστικά ε, αφορούν 45.000 εκτάρια. Πρέπει να δούμε δηλαδή ότι ε, ανάμεσα στα, ε, ποσά, στα εκτάρια που ανακοινώνονται και στα εκτάρια που τελικά χρησιμοποιούνται υπάρχει συνήθως ένα, μια μεγάλη διαφορά. Το 2012 υπήρξε μία μελέτη που κατέγραψε όλες τις επενδύσεις που έγιναν από το 2008 μέχρι το 2009 που είχαν δρομολογηθεί, τέλος πάντων δρομολογούνταν τότε, 2008 και 2009 σε 81 χώρες, 464 ε, προγράμματα, 46 ε, εκατομμύρια εκτάρια, εκ των οποίων τα δύο τρίτα αφορούσαν την ε, Αφρική. 35% ήταν ακόμη εκμετάλλευση, ήταν ακόμη όχι ακόμη υποεκμετάλλευση. 18% των 46 εκατομμυρίων εκταρίων είχαν εγκριθεί από τις εθνικές αρχές, αλλά οι εργασίες εκμετάλλευσης δεν είχαν ακόμη ξεκινήσει. 30% των γεών ε, ήταν σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και 22% των γεών ήταν ε, πράγματι υποεκμετάλλευση. Σε μία μελέτη που εμφανίστηκε το 2011, το International Loan Coalition ε, καταγράφει 203 εκατομμύρια εκτάρια ε, αντικείμενο ανταλλαγή ε, μέχρι το 2010, το 2001 μέχρι το 2010. Από τα 203 εκατομμύρια εκτάρια μπόρεσε μόνο 71 εκατομμύρια να ελέγξει 78% εκ των οποίων είναι γεωργικής παραγωγής και τα υπόλοιπα ήταν ε, ε, ε, τουριστικές εγκαταστάσεις ή ορυχεία. Είναι απλώς νούμερα, αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η πλαισίωση στο μυαλό μας με τα νούμερα αυτά. Το International Loan Coalition λέει ότι υπάρχει μία επιβράδυνση τα τελευταία χρόνια, όμως παραμένει σημαντικό το φαινόμενο και ότι δεν είναι δυνατόν ε, να συνεχίσει κάτι τέτοιο. Ε, τα βιοκαύσιμα αυξάνεται η ζήτησή τους, ε, άλλωστε αναφέρθηκε και σήμερα το πρωί, αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, έκρηξη των αστικών κέντρων, επίσης εμφάνιση πληθυσμών στις αναδυόμενες χώρες και στις αναπτυσσόμενες χώρες ε, μιας μέσης τάξης, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν τρώμε το ίδιο πράγμα. Όταν είμαστε ε, φτωχοί δεν τρώμε το ίδιο πράγμα που τρώμε όταν είμαστε σε μια μεσαία τάξη. Αυτό σημαίνει λοιπόν μια διατροφική μετάβαση και πρέπει να σας επιστήσω την προσοχή σε αυτό το θέμα. Γιατί υπάρχει μια διατροφή όλο και περισσότερο με κρέας και όλο και περισσότερο, με όλο και περισσότερη ποικιλία. Όμως φαίνεται επίσης ότι η κατανάλωση του, κρέωτας, του κρέατος ε, σημαίνει περισσότερη χρήση ε, χώρου και περισσότερη χρήση ζώων. Δηλαδή ε, τα ζώα και αυτά προκειμένου να βοσκήσουν, για παράδειγμα, χρησιμοποιούν περισσότερο χώρο. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν μια τυπολογία, αλλιώ δεν βλέπουμε πόσο περίπλοκο είναι το θέμα. Τι γίνεται με τι άμεσε επενδύσει στην υποσαχάρια Αφρική. Πρώτον, υπάρχουν χώρε οι οποίε θέλουν να εξασφαλίσουν ε, την ε, διατροφική του προμήθεια σε μεγάλο χρονικό διάστημα, μακροπρόθεσμα. Σαουδική Αραβία, Κίνα, χώρε του Περσικού κόλπου, Λιβύη πριν ε, από την πτώση του Μαμάρ Καντάφη, ήταν σε μια στρατηγική μετεγκατάσταση τη διατροφική του παραγωγή, δηλαδή έκαναν σε αφρικανικές χώρες και το έβλεπαν αυτό ως λύση για την ε, κακή διατροφή, ε, ε, τον υποσυτισμό των πληθυσμών τους, οι πληθυσμοί τους οποίους πλήττει αυτό είναι οι, οι πληθυσμοί των οποίων οι χώρες κάνουν τις επενδύσεις. Έχουμε την Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, την Ινδία, την Κίνα και αυτοί προβαίνουν σε αυτές τις στρατηγικές ε, ε, γιατί όλο και περισσότερο ακριβό είναι για τις φακές, για παράδειγμα, που παράγονται στην Ινδία. Είναι όλο και πιο ακριβές οι φακές στην Ινδία και επομένως ε, μετεγκαθιστούν την παραγωγή τους στις ε, αφρικανικές χώρες γιατί το κόστος παραγωγής είναι πολύ χαμηλότερο. Δεύτερο είδος ε, εταίρων είναι η παραγωγή βιοκαυσίμων. Τα βιοκαύσιμα είναι πάρα πολύ παρόντα σε όλη αυτή τη διαδικασία και σε αυτό το φαινόμενο όταν παρουσιάζονται οι επενδύσεις ε, στη γεωργία ως λύση στο διατροφικό ε, ε, πρόβλημα, στο επιστητικό πρόβλημα, δεν σημαίνει ότι αυτό θα θρέψει τα στόματα βέβαια, γιατί βλέπετε τι, τι προβλήματα δημιουργεί. Επίσης, συνταξιοδοτικά ταμεία αρχίζουν να ενδιαφέρονται για αυτή την περιοχή και για τις επιχειρήσεις που επενδύουν ε, στις ε, ε, γέες αυτές. Είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον αυτό, γιατί τα συνταξιδοτικά ταμεία σκέφτονται πολύ απλά. Είναι ένας σημαντικός τομέας, αυξάνεται ο πληθυσμός της γης, θα αυξηθεί και η τιμή της γης, επομένως πολύ καλό είναι να επενδύσουμε στις συγκεκριμένες χώρες και αυτό δημιουργεί ένα επιπλέον φόρτο, ένα επιπλέον βάρος. Και έχουμε επίση και τα αφρικά κράτη, τα οποία τα ξεχνάμε, αλλά είναι οι πρώτοι εταίροι. Θέλουν ε, να υποδεχθούν ε, ξένες άμεσες επενδύσεις ε, στα εδάφη τους, γιατί αυξάνει το ΑΕΠ τους, γιατί πιστεύουν ότι θα, θα λύσει κάποια προβλήματα, το εμπορικό ισοζύγιο και πολλά άλλα πράγματα. Οι, ε, τα, αφρικανικές χώρες, 20 σήμερα, ε, είναι προορισμός τέτοιου είδων επενδύσεων ε, ή ψάχνουν τις επενδύσεις και γίνεται ένα κοινωνικό dumping και φορολογικό για να υπάρξει η καλύτερη προσφορά στους επενδυτές. Δηλαδή, ε, δεν θα σας ε, ζαλίσουμε και με όλα αυτά τα θέματα της εγγύου ιδιοκτησίας, θα βρούμε διαθέσιμες γεές, ενώ στην ουσία δεν είναι καθόλου διαθέσιμες αυτές οι γεές και τα αφρικανικά κράτη είναι στο επίκεντρο αυτής της δυναμικής. Υπάρχει και ένα τελευταίο είδος ε, ε, εταίρου που είναι οι διεθνείς οργανώσεις, μιλήσαμε για την Παγκόσμια Τράπεζα που το ευνοεί. Αυτό λέει ας πούμε ότι ε, κάθε ξένη άμεση επένδυση καλή είναι στις αφρικανικές χώρες. είναι καλό οι χώρες αυτές να έχουν άμεσες επενδύσεις ξένες. Όσον αφορά τώρα τις συνέπειες, πρέπει, ειδικά σε αυτό το τομέα, να δούμε τις λεπτομέρειες, γιατί ο διάβολος εκεί κρύβεται, στις λεπτομέρειες. Δύο είδη υπεχειρημάτων υπάρχουν. Κάποιοι λένε ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι ε, εκφύσεως κακές, ε, ότι είναι, ομά, ότι είναι η μεταμφίεση μιας ε, νέας απεικιοκρατίας και από την άλλη υπάρχει το επιχείρημα ότι όχι αυτές οι επενδύσεις εκφύσεως είναι πολύ καλές για την απασχόληση, θα ενθαρρύνει την γεωργία, θα δώσει τη δυνατότητα δημιουργίας υποδομών κλπ. Προσπαθούμε να βρούμε μια γραμμή που μπορεί να συγκεράσει αυτά τα δύο άκρα. Για μένα το βασικό ζήτημα έγκυται στη δυνατότητα των κρατών να πλαισιώνουν και να συνοδεύουν αυτές τις επενδύσεις. Εκεί έγκυται το ουσιαστικό ζήτημα. Υπάρχει μια μελέτη η οποία εκπονήθηκε από τον Λορέντζο Κοτούλα, έναν ερευνητή για το International Institute ε, of Environment and Development και από το ΦΑΟ. Το 2009 πήγαν σε 8 αφρικανικές χώρες, προσπάθησαν να βρουν αυτά τα συμβόλαια τα περιβόητα, τα μελέτησαν και το συμπέρασμα τους ήταν αρκετά απεσιόδοξο. Πρώτον, υπάρχει μια δυσκολία πολύ σημαντική ε, πρόσβαση στα συμβόλαια αυτά. Δεύτερον, όταν είχαν την πρόσβαση αυτή στα συμβόλαια, τους εξέπλησε και τους τρομοκράτησε το γεγονός ε, ότι μερικές φορές μιλάμε για δεκάδες και εκατοντάδες εκτάρια που νοικιάζονταν ε, για ε, δεκαετίες ολόκληρες μέσα σε τέσσερις σελίδες. Όταν μιλάω βέβαια για το μέγεθος των συμβολέων αυτών, καταλαβαίνετε τι θα πει για τις λεπτομέρειες της, των συμβάσεων αυτών. Ε, και μάλιστα η ζώνη των επενδύσεων δεν ήταν καν καταγεγραμμένη στο κτηματολόγιο. Λέγαμε ας πούμε ότι ήταν ε, τάδε αριθμό εκταρίων, αλλά δεν είχε κάνει καν το κράτος την προσπάθεια να εντοπίσει που βρίσκονται αυτές οι γέ που είχε σκοπό να μισθώσει. Επέστησε την ε, προσοχή και σε ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα, ότι η διαδικασία ε, διαπραγμάτευσης μεταξύ των κρατών και των ε, εταιριών ε, επενδυτών είναι συνήθως πολύ κεντρική από την, πλευράς, από την πλευρά των κρατών, των κρατών των Αφρικανικών. Ο ίδιος συχνά ο, πρό, πρόεδρος ή ο πρωθυπουργός το κάνει. υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες τις οποίες θα έπρεπε να έρθει, με τις οποίες θα έπρεπε να έρθει σε επαφή η θήνους αρχή δεν το έκανε. Οι επενδύσεις δεν ε, πλαισιώνονται λοιπόν καλά από τις αρμόδιες αρχές του κράτους. Ε, μόνο οι προεδρίες ε, αναλαμβάνουν τη διαπραγμάτευση και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν ε, σημαίνει λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ καλό το οικονομικό αποτέλεσμα των συμβολέων αυτών. Είναι πολύ λίγο δεσμευτικέ. Αν ναι, θα κάνουμε κέντρα υγεία, θα κάνουμε υποδομέ, ε, ε, θα ενισχύσουμε την τοπική γεωργία. Αλλά δεν υπάρχει κανένα απολύτω αριθμό που αναφέρεται. Είναι πάρα πολύ αόριστα όλα αυτά και δεν είναι καθόλου δεσμευτικέ. Είναι απλώ δηλώσει προθέσεων το κράτος ε, δεν δεσμεύει σε τίποτα τον επενδυτή. Άρα, εν κατακλείδη, από τις διάφορες μελέτες που έγιναν, ως προς επιπτώσεις των επενδύσεων, βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που ήταν θύματα αυτών των επενδύσεων. οι μικροαγρότες, οι φτωχοί αγρότες των ε, αγροτικών περιοχών που δεν βρίσκονται κοντά στην ε, κεντρική εξουσία. Η δεύτερη κατηγορία, και αυτό προελέχθη, είναι οι κτηνοτρόφοι, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για αυτούς, και έχουν δικαίωμα χρήσης γεών μέσα στα πλαίσια όμως μιας γενικότερης επισφάλειας δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν καθαρά αγροτεμάχια. Και η τρίτη κατηγορία είναι οι γυναίκες. Σε πολλές αφρικανικές χώρες, όπως και στη δική μου χώρα, υπάρχουν γυναίκες επικεφαλής γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ζουν κάτω από συνθήκες επισφάλειας. Και γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλές φορές αυτές οι συμβάσεις στην καλύτερη των περιπτώσεων οδηγούν σε ένα κτηματολόγιο και ορίζουν την εκμετάλλευση της γης, αλλά δεν μιλάν για τους κινδύνους που ελοχεύουν. Υπάρχει πρόβλημα προσβασιμότητα στη γη, αλλά φανταστείτε μία επιχείρηση από την Ινδία η οποία επενδύει στην Αιθιοπία και θέλει να προβεί σε καλλιέργεια λουλουδιών. Δεν έχει πρόσβαση στο νερό. Πού θα πρέπει, θα πρέπει να βασιστεί στον υδροφόρο ορίζοντα που προϋπάρχει. Τι θα κάνει, θα κάνει γεωτρήσεις, γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη από κοινού τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους. Να σκεφτόμαστε, να σκεφτόμαστε τα δικαιώματα επί της γης, την επιφάνεια των καλλιεργήσιμων γεών, τις αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης ή απαλωτρίωσης, αλλά και την ε, πρόσβαση στο, στον υδροφόρο ορίζοντα. Η Αφρικανή παραγωγή και κτηνοτρόφοι χρειάζονται ασφάλεια με την απλούστευση ιδιοκτησιακού καθεστώτος. γιατί οι γεωργοί δεν μπορούν να προβούν σε επενδύσεις αν δεν είναι σίγουροι ότι θα έχουν τη γη τους σε 10 χρόνια. Είναι τόσο απλό. Ένας ε, Αφρικανός γεωργός είναι ένας όμο και αν δεν γνωρίζει ότι μπορεί να κρατήσει τη γη του, γιατί να κάνει επενδύσεις. Δηλαδή, αν σας δίναν γη για να οικοδομήσετε και σας λέγανε ότι αυτή τη γη την έχετε για 20 χρόνια, θα χτίζατε? Όχι βέβαια. Δεύτερον, οι αγρότες και ιδιαίτερα οι μικρογεωργοί χρειάζονται συνοδευτικά μέτρα. Και εδώ επανέρχομαι στην γεωργική πολιτική των αφρικανικών χωρών. Χρειάζονται λιπάσματα, σπόρους, στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Το κράτος θα πρέπει να διοργανώνει τη συγκομιδή εκεί που δεν μπορεί να το κάνει ο ιδιωτικός τομέας. Αλλά αυτό γίνεται 15-20 μέρες αργότερα και δυστυχώς έχουμε παραγωγή η οποία σαπίζει στην άκρη του δρόμου. Αγροτική πολιτική σημαίνει μίζωνα επενδυτική πορεία του κράτους. Και επίσης οι μικροαγρότες θα πρέπει να έχουν πιστώσεις διαφορετικά. Αυτοί που έχουν μικρά αγροτεμάχια χωρίς ασφάλεια τι θα κάνουν. Δεν επενδύουν στα δικά τους αγροτεμάχια αλλά στις πολυδραστηριότητες. Δηλαδή μεταφέρουν, γίνονται έμποροι, βιοτέχνες κατά της απόδοσης της γης. Και αυτό το βλέπουμε στην υποσαχάρια Αφρική τα 30 επόμενα χρόνια η γεωργία θα πρέπει να αυξήσει την απόδοσή της και αυτό μπορεί να γίνει μόνο υπό τους όρους που προαναφέραμε. Και το τελευταίο ζήτημα αφορά το παραδοσιακό δίκαιο. Όπως είπε και ο κύριος Αρισού, το εθνικό δίκαιο πολλές φορές μπορεί να υπερσκελιστεί και στο Σαχέλ, στη Δυτική Αφρική, υπάρχει μία κάστα επενδύσεων και επιχειρήσεων. Ποιος έχει πρόσβαση στη γη, οι μεγαλογεοκτήμονες και όχι οι φορολογούμενοι, γιατί αυτό θέτει ένα αμφιβόλο το εθιμικό δίκαιο. Αλλά θα πρέπει να το δούμε και από την καλή και από την κακή πλευρά. Άρα τα ζητήματα που μας απασχόλησαν σήμερα είναι πολύ πιο ευρεία από το πετρέλαιο, τα διαμάντια και ούτω καθεξής. Γιατί πάντα υπάρχει μία διάσταση εγγύου ιδιοκτησίας ακόμα και σε περίπτωση σειράξεων στην ακτή του ελεφαντοστού το βλέπουμε αυτό, αλλά θα μπορούσαμε να δώσουμε πληθώρα παραδειγμάτων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε. Έχουμε μερικά λεπτά για τυχόν ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής μας, τους συναδέλφους. Έχετε καμία ερώτηση, παρακαλώ. Ρικάρντο, Φίλιπ. Ναι, Σκέψη περισσότερο. Είναι, δεν είναι ερώτηση. Μετά από τις παρεμβάσεις και των δύο πανελίστ. Όπως είπε και ο κύριος Κασμάρ, υπάρχει ένα θέμα εμπιστοσύνης, πολύπτυχο. Θα πρέπει να βρούμε μία απαρχή λύσεων. Κάτι που θα έπρεπε να έχουμε επιλύσει εδώ και δέκα 15 χρόνια και κάτι το οποίο δεν μας απασχολεί τόσο όσο θα έπρεπε, ούτε και σήμερα, είναι ότι η γη αποτελεί αντικείμενο κερδοσκοπίας, βρίσκεται στα χέρια πολύ λίγων και θα μας απασχολήσει και σε αυτή την Επιτροπή. Σε άλλες περιστάσεις Μιλήσαμε για άμεσες λύσεις πολλές φορές για να προωθήσουμε μία αναπτυξιακή πολιτική, να ορίσουμε την πολιτική αυτή ανάπτυξης με βάση συγκεκριμένες προτάσεις. Οι αφρικανικές χώρες θα βρουν τη λύση. Εμείς δεν μπορούμε παρά να συνεργαστούμε με αυτή την Ήπειρο. Δυσεπίλητο, δεν λέω, αλλά θα πρέπει να θέσουμε σωρία ερωτημάτων έτσι ώστε να εκινήσουμε αυτή τη διαδικασία και τη στιγμή που έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τις αφρικανικές χώρες στο μέτρο του δυνατού. Να εκινήσουμε μηχανισμούς στις αφρικανικές χώρες. Είναι δύσκολη η κατάσταση, πολλές φορές ε, δεν υπάρχει δυνατότητα επίλυσης ε, ζητημάτων. Πολλές πολυεθνικές διαθέτουν γη, όπως είπε και η κυρία Στίφλερ και η πρόεδρος και στην Ινδία και στη Λατινική Αμερική και στην Αφρική. Όπως είπε και ο κύριος Σέφερ, στην Ινδία όταν βρίσκεται μια λύση μπορεί κανείς τουλάχιστον να εργαστεί πάνω σε αυτή τη γη. Γι' αυτό θα πρέπει να διανοίξουμε αυτή τη δυνατότητα και σε άλλες χώρες της Αφρικής. Μαζί με αυτά που είπε, μου, είπα, που είπαν η κυρία Αντίλ και Νουρισάντ. Έχουμε θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν και στο μέλλον. Θα διονγκωθούν στο μέλλον εάν δεν δώσουμε μία λύση τώρα. Γι' αυτό θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε και να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε αυτή τη συζήτηση και να απασχολήσει βεβαίως και τους επιτρόπους μας. Πρόκειται για μια κατάσταση η οποία καρκινοβατεί κάπως. Δεν είμαι αρνητικός, θέλω να είμαι και ε, αισιόδοξος αλλά και ρεαλιστής σύναμα. Πολλές φορές δεν υπάρχει πολιτική θέληση. Κάτι το οποίο έχει σχέση και με άλλα ζητήματα, όπως η κατάσταση διαφθοράς και πολιτικής αστάθειας σε, όλες, σε πολλές χώρες. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ευχαριστώ. Πολύ σκόπιμο το σχόλιο, ήταν σχόλιο και όχι ερώτηση. Αν θέλετε μπορείτε να ε, ε, λάβετε το λόγο. Φιλίπ Κατσμάρκ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μίλησα με το συνάδελφό μας, τον κύριο Ντέβα, ο οποίος είπε, πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να μιλήσουμε μόνο για την καταπολέμηση της φτώχειας, αλλά και για την αύξηση ε, της ευημερίας ή αν θέλετε ακόμα και της περιουσίας. Ε, αυτό το θέμα το συζητούμε πάρα πολλά χρόνια. Στην αρχή είχαμε το κίνητρο του κυρίου Βισότο να νομιμοποιήσουμε, να βρούμε δηλαδή τη νομική βάση για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Ε, η έκθεση που είχε γίνει τότε ε, κατέληγε σε ορισμένα συμπεράσματα ε, τα οποία όμως σήμερα δεν είναι τόσο σωστά όπως τότε όταν συντάχθηκε είδαμε τώρα ότι έχει επικρατήσει το εμπορικό μοντέλο ενώ εμείς θέλαμε να ενισχύσουμε την, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Έχουμε έναν κανόνα σε αυτό το σώμα, ε, σύντομη ομιλία, να είστε κάπως σύντομος. Ναι, κοιτάξτε, λέει ο κύριο Σέφερ, Βεβαίως ε, πρέπει να αυξήσουμε και να ενισχύσουμε και να διασφαλίσουμε την ευημερία, αλλά να τους δώσουμε τα μέσα, τα εργαλεία, να το επιτύχουν αυτό. Καταρχάς αναγνώριση οποιονδήποτε τίτλων που υπάρχουν. Ε, εμάς βεβαίως οι διοκτησίες που έχουμε έχουν δημιουργηθεί κατά καιρού σε χώρες της δύση ε, και εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Όμως δεν μιλάμε γι' αυτό. Ε, στις χώρες που μας ενδιαφέρουν πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε την πολιτική βούληση. Και αυτή δεν είναι εξασφαλισμένη, διότι πολλές φορές βλέπουμε τα χρήματα να πηγαίνουν στις τσέπες των γραφειοκρατών ή των αρμοδίων, αντί στους δικαιούχους. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν μπορούμε να την αρνηθούμε. Δύο σημεία που θα απαντήσουν νομίζω στις ερωτήσεις που ετέθησαν. Το πρώτο είναι το εξής. Υπάρχει, δεν ε, είπα πολλά γι' αυτό, ξένες ή εθνικές επενδύσεις που έχουν ε, θετική συνέπεια στην ε, γεωργία. Είναι συνήθως μικρότερης εμβέλειας και γι' αυτό μιλάμε λιγότερο για αυτές. Υπάρχουν όμως πολλά παραδείγματα και αναφέρομαι κυρίως σε εταιρείες Κένιας, ε, που καλλιεργούν λουλούδια ε, και γύρω από τη ζώνη όπου υπάρχουν οι επενδύσεις αυτές ε, πάει καλύτερα η κατάσταση γιατί χρησιμοποιούν όλη την επένδυση αυτή προκειμένου να καλλιεργούν λουλούδια. Όλο και περισσότερες δηλαδή καλλιεργητές λουδιών υπάρχουν. Οπότε είναι ουσιαστικά κάποιοι μοχλοί ανάπτυξης οι εθνικές, ε, όλες οι εθνικές και ξένες επενδύσεις δεν είναι υποχρεωτικά κακές, απλώς όταν κοιτούμε τις λεπτομέρειες είναι μικρότερες, ε, αφορούν ε, κάποιες εκατοντάδες ή χιλιάδες εκτάρια. Για το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να θέσω για τη Σενεγάλη και τον Υπουργό Γεωργών, Γεωργίας. Ε, είχα κάνει ένα, μια μελέτη για το θέμα αυτό. Είχα πάει και είχα συναντήσει εμπειρογνώμονες ε, Σενεγαλέζους ε, και άλλους εμπειρογνώμονες για τη Γεωργία. Μου είχαν πει δύο πράγματα. Το Υπουργείο ήταν θύμα στη Σενεγάλη, όπως και, πολλέ, και πολλά άλλα Υπουργεία στη Σενεγάλη ή αλλού, πολιτικής ε, δημοσιονομικών περικοπών, ε, περιορισμών τέλος πάντων, ε, όπως από την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το, τη δεκαετία του 1990 υπήρξε ένα πάγωμα μισθών, πάγωμα προσλήψεων και οι συνέπειε είναι ότι σήμερα η Σενεγάλη πληρώνει ακόμη το, τι, το τίμημα. Ένα απλό παράδειγμα είναι η Σενεγάλη. υπάρχει μια, ένα τεράστιο κενό ε, στις προσλήψεις. Υπάρχουν λοιπόν προσλήψεις που έγιναν πολύ τελευταία στιγμή. Υπήρχε προβλήματα, υπήρχαν προβλήματα προσλήψεων για 15-20 χρόνια περίπου. Παράλληλα, επειδή πάγωσαν οι μισθοί, μερικά από τα καλύτερα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας ε, ε, έφυγαν, ε, πήγαν σε μη κυβερνητικέ οργανώσει, σε ιδιωτικό τομέα, όπου ήταν καλύτεροι μισθοί βεβαίω. Και να σα πω την αλήθεια, εγώ δεν ε, θα του λιθοβολήσω πρώτος. πολύ σκληρή πολιτική λοιπόν, ε, η οποία σκοπό είχε να, να μειώσει τις δαπάνες των χωρών και αυτό σημαίνει ότι, ότι μπλοκαρίστηκε και η δυνατότητα της χώρας να βασιστεί στη δική της ε, οικονομία. Ε, ένας μεγάλος εμπειρογνώμονας για τα θέματα της ενεγαλέζικης γεωργίας μου είχε πει τότε ότι ούτε το ίδιο το Υπουργείο γνώριζε πολύ καλά τι συνέβαινε σε ολόκληρη την ε, επικράτεια της Σενεγάλης. Ε, πρέπει λοιπόν να νοικοδομήσουμε τα κράτη και αυτό πρέπει να προκύψει από τα ίδια τα κράτη. Δεν είναι δυνατόν να είναι απλώς ε, ξένοι εταίροι αυτοί που θέλουν να επιβάλλουν την ανοικοδόμηση αυτή. Μπορούν να υποστηρίξουν και το κάνουν ήδη σε κάποιο βαθμό τη δυνατότητα των κρατών μελών ε, να ανοικοδομήσουν τις γεωργικές τους πολιτικές. Σχεδόν ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Τώρα θα πάμε από την Πράγα, από τη δική μου χώρα, στο Δουβλίνο, στον συνάδελφό μου. Ευχαριστώ πολύ και σας καλωσορίζω όλους. Δεν θέλω να επαναλάβω τα ίδια λεχθέντα. Θα κάνω μερικές παρατηρήσεις. Καταρχάς, από πλευράς του δικού μου κόμματος, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι νόμιμοι τίτλοι, αν υπάρχουν, μπορεί να επιτρέψουν στους δικαιούχους να δανειστούν, άρα και να επενδύσουν. Γι' αυτό λοιπόν η διασφάλιση ε, της ιδιοκτησίας είναι το πιο σημαντικό δεν μιλούμε, όταν μιλάμε για δικαιώματα ιδιοκτησίας, δεν μιλάμε μόνο για παραγωγούς, για αγρότες και το δικαίωμα ιδιοκτησίας της γης, αλλά αλλάζει όλη του την αντιμετώπιση, όλο το, το, το, το, πώς αισθάνονται. Δηλαδή πολλές φορές απαλλάσσονται από το φόβο που έχουν για το, την εξασφάλιση του μέλλοντός τους από τη στιγμή που έχουν νόμιμους τίτλους. Το λέω αυτό από προσωπική εμπειρία γιατί ξέρω παρόμοιες περιπτώσεις στην Ιρλανδία. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο προσωπικά δικαιώματα που πρέπει να εξασφαλίσουμε αλλά είναι και δικαιώματα της κοινωνίας. Η Παγκόσμια Τράπεζα σε μια έκθεση του 2003 σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φτώχειας στον αναπτυσσόμενο κόσμο, ανέφερε τρεις, ε, τρία σημαντικά, τρεις σημαντικές συνέπειες που μπορεί να έχει η εξασφάλιση των γεών. Πρώτον, ναι, την αύξηση της παραγωγής, διότι δεν θα χάνουν τόσο χρόνο οι ιδιοκτήτες με τη γραφειοκρατία. Δεύτερον, η οι τίτλοι και η διασφάλιση των γεών βεβαίως ε, βοηθούν την παραγωγή, άρα μειώνουν τη φτώχεια. Και τρίτον, βοηθούν την κοινωνική ανάπτυξη ολόκληρων κοινοτήτων. Δηλαδή έχουν και κοινωνικές επιπτώσεις. Πέραν αυτού έχουν υλικά ωφέλη ιδιαίτερα για τις γυναίκες, οι οποίες πολλές φορές είναι ή μικροκαλλιεργητές αυτών των γεών ε, και αυξάνουν επίσης και τη δυνατότητα επιμόρφωσης των παιδιών τους και δι των κοριτσιών. Ε, είναι μία ακόμα μεγάλη, μία προτεραιότητα η καταπολέμηση της φτώχειας. Και εάν δεν διατηρήσουμε αυτό το θέμα ε, ως προτεραιότητα, τότε θα το χάσουμε, θα, θα χαθεί μέσα στη σκόνη τόσων άλλων προβλημάτων. Στο τέλος ε, του Παγκοσμίου Πολέμου είχαμε 44 της χιλής παιδικής θνησιμότητας στην Ιρλανδία. 44 της χιλής. Τώρα έχουμε τη χαμηλότερη παιδική θνησιμότητα σε ολόκληρο τον αναπτυγμένο κόσμο. Στον αναπτυσσόμενο κόσμο είναι 68 της χιλής. Είναι ένα τρομακτικό ποσοστό αυτό, ε, διότι αντιλαμβάνεστε τον αριθμό των νεογνών που πεθαίνουν ε, λόγω της ένδυας και των ελλείψεων. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τον αναπτυσσόμενο κόσμο, όχι μόνο προσφέροντας προγράμματα και πιστώσεις, αλλά προσφέροντας και την εμπειρία μας. Πολλοί από τον αναπτυσσόμενο κόσμο λένε, ισχυρίζονται ότι οι Ευρωπαίοι δεν καταλαβαίνουν. Εγώ ε, έχω αντίρρηση σε αυτή την προσέγγιση. Κοιτάξτε τη δική μου χώρα, κοιτάξτε τη δική μου χώρα και τι έγινε εκεί στην ιστορία της. Από το 1922 είναι διαιρεμένη η Ιρλανδία. Είχαμε μία ε, αγροτική κοινωνία, ήταν αγροτική οικονομία, όπου οι μεγάλοι γεωκτήμονες ήταν απόντες. Και ε, τα, οι τα χωράφια ήταν πάρα πολύ μικρά. Χρησιμοποιούσαν επίσης ε, το μοντέλο της Βρετανίας. Και ε, σιγά σιγά εκμεταλλεύτηκαν αυτές τις γέες ε, στην Βόρειο Ιρλανδία, όπου βεβαίως είχαν την μεγάλη ε, επιρροή από την ε, Βρετανία, από το Ηνωμένο Βασίλειο και συνεχεία βιομηχανοποιήθηκαν ο Βοράς ενώ ο Νότοες έμεινε κολλημένος στην παραγωγή των βασικών ειδών τροφίμων, ας πούμε, για επιβίωση και υπέστη μετά τις γνωστές καταστροφές. Έχουμε, λοιπόν, υπουργό Ιρλανδικών γεών. Ακόμα όταν ήμουν εγώ βουλευτής εθνικός στην Ιρλανδία, είχαμε Επιτροπή Γεών και Υπουργό Γεών. Και ε, πολλά κτήματα αγοράστηκαν τότε από το κράτος, απαλωτριώθηκαν δηλαδή και αγοράστηκαν και κατανεμήθηκαν στους μικροπαραγωγούς προς καλλιέργεια. Ε, η δημοκρατία της Ιρλανδίας άνοιξε ε, ε, ε, τις πόρτες βεβαίως όταν εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγιναν μεταρρυθμίσεις και στην νομοθεσία πολύ πριν από την κυβέρνηση της κυρίας Στάτσερ η οποία είχε πει ότι δεν υπάρχει κοινωνία, υπάρχει μόνο άτομο το άτομο. Λοιπόν, αν, άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα στην Ιρλανδία, χωρίς να αλλάξουμε βεβαίως τον τρόπο που ψηφίζει ο κόσμος. Ήταν ελεύθεροι να ψηφίσουν το ένα ή το άλλο κόμμα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι άνθρωποι είναι ήδη, είτε ζουν στον τρίτο κόσμο, στον αναπτυσσόμενο, στον ανεπτυγμένο, στον πρώτο, έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες αυτές πρέπει να τις εκμεταλλευτούν και η Παγκόσμια Τράπεζα στην έκθεσή της έχει πολύ δίκιο πρέπει αυτές οι τρεις μεγάλες αλλαγές να γίνουν και μπορούν να γίνουν. Όσον αφορά τώρα την νόμιμη, τους νόμιμους τίτλους, την νόμιμη ιδιοκτησία, δημιουργούμε πάρα πολλά εμπόδια στην απόδειξη της νομιμότητας. Ε, παραδείγματος χάρη τα προβλήματα που είχαμε με τη Σιλάνκα. όταν έγινε το τσουνάμι, όταν έγιναν οι τεράστιες πλημμύρες και οι καταστροφές και χάθηκαν οι φράχτες, χάθηκε δεν μπορούσαν να αποδείξουν τα όρια της ιδιοκτησίας. Ε, έχουμε τώρα δορυφορικές ε, τεχνικές διευκολύνσεις, παραδείγματος χάρη τις έχουμε χρησιμοποιήσει και στην Ευρώπη και αλλού. Μέσω δορυφόρων μπορεί να ε, αποδειχθούν ο διαχωρισμό των γεών, η χαρτογράφηση δηλαδή των γεών, για να βοηθήσει ας πούμε στην εδραίωση των τίτλων, κλιματολογία κλπ. Να μην ξεχνάμε λοιπόν και τη σύγχρονη τεχνολογία την οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Βεβαίω, ε, στο παρελθόν οι διαδικασίες ήταν πάρα πολύ αργές και πρέπει να βρούμε μέσα να ξεπεράσουμε αυτή την αργοπορία, αυτή την ε, καθυστέρηση. Είτε μιλούμε για μία μικρή έκταση, για μία μικρή παραγωγική μονάδα, πρέπει να προσφέρουμε κίνητρα ε, στους ενδιαφερόμενους εμάς, στους πολιτικούς μας αρέσει να ελέγχουμε κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής. Εγώ είμαι χριστιανοδημοκράτης, δεν, είμαι, δεν θεωρώ τον εαυτό μου ούτε υπερσυντηρητικό ούτε σοσιαλιστή, είμαι κάπου στη μέση. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να μεταφερθεί η δύναμη από το κράτος, από τον κρατισμό δηλαδή, ε, στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι ε, μπορούν να, πάρουν ε, αποφάσεις για τη ζωή τους και είναι υπεύθυνοι. Ε, ε, ε, με μεγάλη χαρά λοιπόν θα ήθελα να παρουσιάσω τον Bernard Ray και χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι εδώ πρόσωπος της Κομισιόν, διότι υπάρχει το δυναμικό της αλλαγής. Υπάρχει το δυναμικό σε όλους τους κόσμους, ανεπτυγμένους και αναπτυσσόμενους. Ναι, βεβαίως επανερχόμαστε στην ίδια συζήτηση όπως είπε ο κ. Σέφερ ε, είμαστε όλοι πολύ άσχολοι, τρέχουμε από εδώ και από εκεί, στην Επιτροπή, στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ανάπτυξης, αλλά στην ημερήσια διάταξη μας αυτό το θέμα υπάρχει, σε όποια επιτροπή και αν είμαστε. Γι' αυτό με μεγάλη χαρά δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Μπέρνα Τρέι, πρόσωπο της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι από την Γενική Διεύθυνση ΕΦΚΟ και ο κύριος Στευνό είναι μαζί μου από την ίδια διεύθυνση που ασχολείται με θέματα εγγύου ιδιοκτησίας. Γι' αυτό το τρίτο πάνελ θα σας κάνω μία παρουσίαση. ως προς τις δράσεις της Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΒΚΟ για θέματα εγγύου ιδιοκτησίας και τις δράσεις οι οποίες είναι και πιο δυναμικές και ενεργές. Ας κάνουμε ένα βήμα πίσω. Το 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές για θέματα εγγύου ιδιοκτησίας. Επρόκειτο για το ότι τονίσαμε τη σημασία των διοικητικών μεταρρυθμίσεων των επικεφαλής υπουργών για να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα εγγύου ιδιοκτησίας, να ορίσουμε τους κανόνες που προϋπήρχαν, έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο υπάρχουν χάσματα και να δούμε και πώς θα μεταφερθεί αυτό το δίκαιο. Και νομίζω ότι... Α, εντάξει, εντάξει. Πανορθώθηκε η διαφάνεια. Το 2011 ξαναείδαμε το χαρτοφυλάκιο της Ντεύκο ως προς την ιδιοκτησία και είδαμε ότι τα πέντε τελευταία χρόνια, μεταξύ 5 και 12 και 11 μάλλον, είχαμε έναν σημαντικό αριθμό θεμάτων σε 37 χώρες που είχαν σχέση με την ιδιοκτησία. Σημαντικό χαρτοφυλάκιο που σχετιζόταν με ρυθμιστικά ζητήματα, νομικό-ρυθμιστικά, διαχείριση των φυσικών πόρων, ιδιαίτερα των δασών, που είναι ένα καθόδε ζήτημα, καθώς και το ρόλο των τοπικών αρχών στη διαδικασία αποκέντρωσης. καθώς και το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην επίλυση των θεμάτων αυτών, καθώς και την διαμεσολάβηση για την επίλυση των διαφορών και τα ανθρώπινα δικαιώματα που συσχετίζονται με το θέμα. Η μεγάλη όμως αλλαγή από τους διεθνείς κύκλους προέρχεται τα τελευταία χρόνια. Μας έρχεται τα τελευταία χρόνια από τη ΦΑΟ δηλαδή κατευθυντήριες γραμμές για μια σωστή διακυβέρνηση των υγειών, της αλίας και των δασικών εκτάσεων. Πρόκειται για μια διαδικασία που ανέλαβε η ΦΑΟ εδώ και 10 χρόνια και που επιταχύνθηκε από το 2009 όταν είδαμε ότι θα πρέπει να συσχετιστεί αυτό το θέμα με την διατροφική ασφάλεια και φτάσαμε σε ένα έγγραφο για την ε, διατροφική ασφάλεια, το CFS, σε επίπεδο ΦΑΟ. Το 2011 ε, υπήρξαν χρηματοδοτήσεις ε, της Κομισιόν και μετά από τρεις κύκλους διαπραγματεύσεων, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετείχε πλήρως, φτάσαμε σε ένα έγγραφο το οποίο ενεκρίθη από την Επιτροπή για τη Διατροφική Ασφάλεια το Μάιο 2011. Και η έγκριση αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών αποτελεί ένα βασικό βήμα για τη διαχείριση των γεών. Το περιεχόμενο των κατευθυντηρίων γραμμών βασίζεται καταρχήν σε μία σειρά αρχών ως προς τη νομιμότητα, την αναγνώριση της νομιμότητας των δικαιωμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των γεών, τη δικαιοσύνη, την επίλυση διαφορών, την αποφυγή διαφθοράς και την απομάκρυνση κινδύνων. Μιλάμε και για θέματα ε, νομικής αναγνώρισης των γεών γιατί μιλήσαμε για τα δικαιώματα στην αλία, στα δάση, στα βοσκοτόπια, να δούμε κατά πόσο είναι θυμικό το δίκαιο ή όχι και το οποίο πρέπει να τηρηθεί. Υπάρχει και το θέμα της μεταφοράς των αγορών, της αγοράς αυτής και της διαχείρισης. Δηλαδή να δούμε πώς οργανώνονται τα κράτη είτε για να διαχειριστούν τις ε, συναλλαγές περιγεών ή πώς φορολογούν, ποιο είναι το φορολογικό καθεστώς. Και αυτό είναι άκρος σημαντικό. Πρόκειται για κατευθυντήριες γραμμές που βρίσκονται σε θελούσια βάση. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε το συμβατικό δίκαιο, αλλά να βοηθήσουμε τις χώρες που θέλουν να προχωρήσουν ως προς βέλτιστες ή χρήστες πρακτικές. Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές αντικατοπτρίζουν μία αλλαγή στον τρόπο σκέψης. Με βάση όλο ένα και διονγκούμενη ζήτηση και μειούμενη προσφορά υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός που αφορά και το προϊόν κάθε αυτό αλλά και τους φυσικούς πόρους. Άρα, θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη διαχείριση. Δηλαδή τους μηχανισμούς που διέπουν τον όλο μηχανισμό. Και το δεύτερο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να προωθήσουμε σωστές και υπεύθυνες πρακτικές και οι πρακτικές αυτές είναι εκείνες που ορίζονται από τις κατευθυντήριες γραμμές. Η ΦΑΟ μετά από την έγκριση αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών έφτασε σε ένα πρόγραμμα δράσης γιατί τι μπορεί να γίνει για να ε, βελτιωθεί αυτή η διαχείριση γεών. Ε, euh, είτε σε επίπεδο κρατών με πλατφόρμες διαβούλευσης γιατί θα πρέπει η κοινωνία των πολιτών να εμπλακεί και να μιλήσουμε για τις σχέσεις κράτους και γεωκτήτη. Να δούμε ποιες είναι οι διαφορές και να δούμε πώς προοδευτικά μπορούμε να φτάσουμε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Πρόκειται για μακροχρόνια διαδικασία βεβαίως. Είχαμε μια σειρά περιφερειακών προτεραιοτήτων, ιδιαίτερα στις αφρικανικές χώρες και ανά τον κόσμο που ανέλαβε η ΦΑΟ για να προωθήσει αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και να δώσει συνέχεια στο θέμα. Μία δεύτερη ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία αφορά το γεγονός ότι ορίστηκε μία διεθνής ε, συμμαχία που αφορά και πολλούς διεθνείς οργανισμούς, χώρες δωρητές και διεθνείς μικιό. Ε, με βάση τις εργασίες της ΦΙΝΤΑ στη Ρώμη εργάστηκε επί μία πενταετία για ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των γεών και υπάρχει ένα σύστημα δεδομένων online για τις μεγάλες ε, συναλλαγές αγοραπολισίες ε, γεών που αναγνωρίζεται διεθνώς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως. Μιλάμε για μια σειρά εγγράφων, γύρω στα χίλια. Και στο πόρταλ, σε αυτή τη διεύθυνση, βλέπετε τις συναλλαγές αυτές. Είναι μια βάση δεδομένων πολύ σημαντική. Ιδιαίτερα αυτή η χαρτογράφηση σας δίνει ανά τον κόσμο να δείτε ποια, είναι η χαρτογράφηση των γεών. Μιλάμε για 30 εκατομμύρια εκτάρια που αφορούν αυτές τις ε, διεθνείς συναλλαγές. Η συμμαχία αυτή προέβη στη σύσταση ενός παρατηρητηρίου και ορισμένες χώρες έχουν ε, καλύτερες πληροφορίες για αυτές ε, τις συναλλαγές. Και όπως ελέγχθη υπάρχουν δυσκολίες, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τι τεκμηρίωση υπάρχει σε επίπεδο Αφρικής, όπου το σύστημα αγεών είναι επίκαιρο, θα πρέπει να μιλήσουμε για μια πρωτοβουλία της Αφρικανικής Ένωσης που υποστηρίξαμε από το 2006, Land Policy Initiative, που οδήγησε σε μία πλαισίωση του θέματος, προωθώντας για όλες τις αφρικανικές χώρες ένα πλαίσιο ύψης της πολιτικής αξίας. Η Υπουργοί Γεωργίας ενέκριναν το 2009 και έτσι η Ήπειρος ξεκίνησε με την εφαρμογή αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών έτσι ώστε να υπάρχουν εξελίξεις ως προς το δίκαιο εγγύου ιδιοκτησίας στην Αφρικανική Ήπειρο. Υπάρχουν και άλλα προγράμματα τα οποία υποστήριξε η Κομισιόν και θα υποστηρίξει στο μέλλον. Μίλησα για τη Διεθνή Συμμαχία για την ε, ιδιοκτησία των γεών που θα προωθηθεί για την επόμενη πενταετία Έχουμε και τις αποφάσεις των G8 για τη διατροφική ασφάλεια. Έχουμε την απόφαση των G8 για τη διατροφική ασφάλεια, όπου εμπλέκονται και οι υγιές, το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Θα πρέπει λοιπόν όλα να είναι συμβατά με αυτές τις δηλώσεις των G8. Και Τέλος θα υποστηρίξουμε την ΦΑΟ για να δοθεί συνέχεια των ε, εθελούσιων κατευθυντηρίων γραμμών ε, τις οποίες προανέφερα. Εδώ βλέπετε τι θα κάνει η ΦΑΟ για την πρόθεση κατευθυντηρίων γραμμών, αξιολόγηση, προώθηση της γνώσης και εταιρικότητας, προώθηση δυναμικού στις χώρες, επιτοπίως καθώς και προώθηση των ε, χρηστών πρακτικών γενικότερα. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται από κοινού με αυτό το θέμα ως προς αυτό το θέμα της εγγύου ιδιοκτησίας. Υπάρχει μια ομάδα εργασίας όπου συμμετέχουν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, συνέρχεται σε τακτά χρονικά δημαστήματα εδώ και μία τριετία για ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων ως προς τη γενικότερη συλλογιστική που μας διέπει για να φτάσουμε σε προγράμματα στήριξης για να εργαστούμε από κοινού με τις χώρες που μπορούν να προβούν σε καινοτόμους πολιτικές και να έχουμε και μία χαρτογράφηση για το τι γίνεται στην Ευρώπη από τα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα. Τέλος, νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το θέμα της γεωκτησίας θα πρέπει να μας απασχολήσει και με στα πλαίσια της διατροφικής ασφάλειας και εξαιτία της επίλυσης διαφορών και σειράξεων ακόμα που έχουν ως αρχέτυπο, ας το πούμε έτσι, προβλήματα για την κατανομή των γεών. Το θέμα της γεωδιακυβέρνησης είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει γενικότερα και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως γνωρίζετε, θα υποστηρίξει τις κατευθυντήριες γραμμές μαζί με την ΦΑΟ. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι χώρες ε, ορίζουν διαφορετικές πολιτικές, πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να γνωρίσουμε ότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις απτές επιτόπιες πραγματικότητες και οι υπηρεσίες μας θα προωθήσουν το ζήτημα για να δούμε τις επιπτώσεις στις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Σας ευχαριστώ. Okay, thank you very much, colleagues. And... Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. <clears throat> Σχόλια. Charles. Ευχαριστώ πολύ. Ένα ερώτημα θα ήθελα να θέσω στον τελευταίο ομιλητή. τι βαθμό αντίστασης ε, βρίσκεται εσείς ότι υπάρχει στις ε, χώρες ε, εταίρους μας. Καλό είναι να υπάρχουν παρατηρητήρια, καλό είναι να υπάρχει αλλαγή και μεταβίβαση τίτλων ιδιοκτησίας κλπ. Αλλά πώς είναι δυνατόν να προχωρήσουμε με τις χώρες εταίρους μας, να εξασφαλίσουμε τη διακυβέρνηση αν εκείνες κάνουν την επιλογή να παραμένουν οι ε, γιες μόνο ε, στην, ε, στην γεωργία. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν θα χρειάζονταν οι χώρες αυτές τους υπόλοιπους. Ποια είναι λοιπόν η κατάσταση, μήπως μπορείτε να μας πείτε, να μας δώσετε μια ιδέα τέλο πάντων για τις δυσκολίες που συναντάτε στην ε, συνομιλία σας με τις χώρες αυτές. Ρικάρντο. Δεν έχω ερώτηση, μία παρατήρηση. Καταρχάς, πιστεύω ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε την ε, Κομισιόν και να συνεχίσει με αυτή την ε, εργασία. Είναι σημαντική από την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μια προτεραιότητα, όπως είπε και ο Σάρλ. Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά τι συμβαίνει, γνωρίζετε την καρδιά του προβλήματος. Ας επιτεθούμε λοιπόν στην καρδιά του προβλήματος και από την Κομισιόν και από το Συμβούλιο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρε, Η Κομισιόν παρακαλώ να απαντήσει ο κύριος Ρέι. Σχέση με το πρώτο ερώτημα για τη δυσκολία ε, του να εργαστεί κανείς στις χώρες εταίρους, εταίρους μας, υπάρχουν διάφορα είδη καταστάσεων. οι χώρες στις οποίες είναι δύσκολο να εργαστεί κανείς και που παρουσιάζουν μια αντίσταση σε σχέση με την ε, αποσαφήνιση της ρύθμισης ε, και της διακυβέρνησης ε, της κατοχής γης. Ε, προσπαθούμε να εργαστούμε σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών για να υπάρξουν πιέσεις και ειδικότερα σε σχέση με την εξαγορά γεών μεγάλου, μεγα, μεγάλων εκτάσεων. είτε τα ELC είτε οι εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές ε, είναι ε, ε, δράσεις τις οποίες προ, προωθούμε προκειμένου να προσχωρούν σε αυτές οι χώρες και προσπαθούμε να έχουμε πλατφόρμες ε, στις οποίες συμμετέχουν και οι κυβερνήτες και οι εκπρόσωποι των γεωργών και η κοινωνία των πολιτών ε, και οι διεθνείς ε, οργανισμοί. Μπορώ να πω και εγώ ορισμένα πράγματα. Δύο οπτικές γωνίες νομίζω, υπάρχουν ε, και είναι στη διάθεση των της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πρώτον, προώθηση μια κοινωνική, μιας κοινωνικής βάσης ε, η οποία να, να ε, ασκεί πίεση και υπάρχει επίσης και εγγραφή στον πολιτικό διάλογο που έχουμε τακτικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση του θέματος της εγγύου ιδιοκτησίας. Συχνά βλέπουμε ότι στον πολιτικό διάλογο είναι ένα ζήτημα το οποίο λιγότερο ε, το προσέχουμε. Χρειάζεται όμως μια ιδιαίτερη προσοχή. Χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή για το θέμα αυτό στις επαφές που έχουμε με τις τρίτες χώρες. Κάρλος. Ναι, ναι, μία παρατήρηση ακόμα. Ένας από τους προηγούμενους ομιλητές μας είπε σαφέστατα ότι σε αυτά τις τακτικές συναντήσεις με, τα, με τους εκπροσώπους των χωρών της Αφρικής ή της Νοτιού Αμερικής δεν διαπιστώνουμε και κανένα μεγάλο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας ή την ασφάλεια των γέων. Μήπως θα πρέπει να συναντηθούμε και να παρακινήσουμε τους αρμόδιους να ξεκινήσει ή να γίνει πιο έντονη η συζήτηση αυτού του θέματος. Θα ήθελα να ξέρω όμως από απόψη συγκεκριμένου αποτελέσματος τι έγινε. Καλό είναι να υπάρχουν περισσότερες συμμαχίες και περισσότερες προσπάθειες, όμως θέλω να μου πείτε τα συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα ποια ήταν ω τώρα. Στη Μαδαγασκάρη ε, προωθήσαμε ένα σύστημα ε, ε, πιστοποιητικών εγγύου ιδιοκτησίας ε, ε, δεκάδες, γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ χρήσιμοποιήσαμε για το σκοπό αυτό ότι να μπορεί κάποιο να πάρει ένα πιστοποιητικό εγγύου ιδιοκτησία ε, βάσει του κτηματολογίου για να μπορεί να πάει σε μια τράπεζα και να πάρει δάνειο. Το κάναμε αυτό σε επίπεδο μικρών ε, γεωργών για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την κατοχή γης, να την, ε, να την εγγυηθούμε είναι ένα τμήμα των 93 προγραμμάτων που έχουμε ε, δρομολογήσει. Ε, προσπαθούμε λοιπόν να δούμε όλα τα συγκεκριμένα ε, προγράμματα που έχουμε στη διάθεσή μας. Ωραία, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας και ευχαριστώ όλους με τις, που, για τις εισηγήσεις τους, τους, τα μέλη μας για τα σχόλιά τους και τους γερμηνείς. Ευχαριστούμε και εμείς. Ε, ξεκινήσουμε ξανά το απόγευμα με την ψηφοφορία για το βραβείο Ζαχάροφ. Θα είναι στο 6Q2, στην αίθουσα 6Q2, ε, στο κτηρίου Q απέναντι, όχι εδώ.